Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Point number one. Σημείο υπαριθμών 1. Έγκριση της ημερησίας διάταξης. Αποουσιάζει ο κύριος Παντσέρη σήμερα, αλλά θα έρθει αύριο. Γι' αυτό και θα αλλάξει η σειρά η έκθεσή του. και ε, αύριο στις 4.45 θα συζητήσουμε τη συστάση, σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 67η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Διαφωνείτε με τα πρακτικά της 28ης ε, Φεβρουαρίου, όχι. Ανακοινώσεις Πρόεδρου θα σας τις κάνω αργότερα, για να μην χάνουμε χρόνο τώρα. Και καλωσόριζω θερμότατα ενώπιόν μας το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Άντερς Φόγκ Ράσμουσεν. Χαίρομαι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σχεδόν τελευταία στιγμή σας το και παραμονές της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο. Χρόνο δεν έχουμε απεριόριστο, άλλη φορά περισσότερο. Να συζητήσουμε τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ πολύ πιο εντατικά ε, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συσφίξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ, πιστεύω. Αλλά ε, του παρόντος είναι σημαντικό που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε να ε, ανταλλάξουμε απόψεις. Έχουμε εκπροσώπους και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, 10 συναδέρφους από 7 Εθνικά Κοινοβούλια. καλωσορίσατε, χαιρόμαστε που είστε νομπέρο μας και θα συζητήσετε κι εσείς μαζί μας με το Γενικό Γραμματέα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε δύσκολη φάση μετασχηματισμού και εμείς στην Ευρώπη ζούμε οικονομική κρίση και είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαζόμαστε περισσότερο και σε θέματα στρατιωτικά και αμυντικά ε, και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας ε, για θέματα όπως είναι επέβαση στη Λιβύη, η κατάσταση στο Αφγανιστάν, η διευρυμένη εντολή της επιχείρησης Αταλάντη. Όλα αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και σας ευχαριστούμε κύριε Γενικέ που εκμεταλλευτήκατε την ευκαιρία αυτή να έρθετε εδώ και να μας ενημερώσετε για τα βασικά σημεία της Συνόδου Κορυφής στο Σικάγο. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Έλμαρ, σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας αποτίσω ένα φόρο τιμής για τη διαρκή σας προσήλωση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Είστε ε, ενεργώς στη συμμετοχή σας ε, στην μεταξέλιξη και τη θεσμική μεταξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε ιδιαίτερα στρατευμένος σε πολιτικές ε, ε, που άπτονται των αμυντικών και εξωτερικών θεμάτων και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, πάντα χαίρομαι όταν επισκέπτομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θα γνωρίζετε ορισμένοι από εσά ότι επί 31 ε, έτη ε, διατέλεσα και εγώ βουλευτής, οπότε αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στο Κοινοβούλιο. Και πάντα είναι καλό και χρήσιμο να θυμίζουμε πόσο ε, κοντά και γεωγραφικά είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ, στην πόλη τούτη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η Ευρώπη έχει λόγο να είναι υπερήφανη. Την περασμένη δεκαετία οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ε, ήταν ο πυρήνας στο Αφγανιστάν ε, βοήθησαν ε, να φύγουν οι περισσότεροι που έφυγαν από τη Λιβύη και βοήθησαν να σταθεροποιηθούν τα Βαλκάνια. Την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη Γεωργία, στα Βαλκάνια και στην Αφρική. Αυτό είναι όντως εντυπωσιακό, όσο και σημαντικό διότι η Ευρώπη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσει στη διαφύλαξη της ασφαλειάς μας. Μπορεί η καιρή που ζούμε να μην είναι η πιο επικίνδυνη στην πρόσφατη ιστορία μας, είναι όμως η πιο περίπλοκη και η πιο απρόβλεπτη. Οι οικονομίες μας ασκούν αφόρητη πίεση στους λαούς και στα δημόσια οικονομικά μας ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλη η κατάσταση και απρόβλεπτη και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή μέχρι και την εμφάνιση και την ανάδυση νέων στρατιωτικών δυνάμεων και νέων απειλών όπως είναι οι επιλές στον κυβερνοχώρο και οι επιθέσεις. Αυτός ο κύκλος πρέπει να τετραγωνιστεί. Έχουμε λιγότερους πόρους στις χώρες μας, αλλά ακόμα μεγάλη βεβαιότητα στον κόσμο. θα πρέπει να εστιαστούμε και στα ε, του οίκου μας, αλλά να μην ε, εθελοτυφλούμε απέναντι σε ένα κόσμο που ε, αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία χώρα από μόνη της, καμία υπερδύναμη και καμία ήπειρος, όσο ισχυρή και να είναι, που να μπορεί από μόνη της ε, και αμέσως να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Τώρα περισσότερο παραποτέ εξαρτώμεθα ένας από τον άλλο για να εξασφαλίσουμε από κοινού ε, την ασφάλειά μας και να διαφυλάξουμε τις κοινέ μας αξίες. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις ε, σχέσεις ασφαλείας που έχουν σημασία. Πάνω από 60 χρόνια η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική έχουν συνεργαστεί στο ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις. Για να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία για να αναπτύξουμε μια Ευρώπη ε, ειρηνική στο σύνολό της και ελεύθερη στο σύνολό της. Σήμερα η ασφάλειά μας δεν μπορεί να ειδωθεί ξεχωριστά από την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτό καμιά φορά σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας και πέραν των συνόρων μας για να είναι ασφαλείς οι πληθυσμοί μας στις χώρες μας. Όπως άλλωστε έχουμε πράξει στο Αφγανιστάν στα νυχτά των ακτών της Σομαλίας και στους εθέρες της Λιβύης. I Γι' αυτό πιστεύω ότι ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των οικονομικών της προβλημάτων η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό της να αναλώνεται σε εσωστρέφεια ή να είναι απορροφημένη μόνο με τα εσωτερικά της. Όταν πρόκειται για ασφάλεια, η μόνη προοπτική που έχει νόημα είναι η παγκόσμια προοπτική. Θα ήθελα όμως να το διευκρινίσω αυτό. Δεν εννοώ ότι αυτόματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει ανά τον κόσμο. Σημαίνει όμως ότι οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να είναι εξωστρεφείς και να είναι σε ετοιμότητα αλλά και ε, να έχουν την προθυμία και την ικανότητα να δρουν από κοινού. Σε συνεργασία με τους Βόρειο-Αμερικανούς ε, συμμάχους μας ε, σε επιχειρήσεις εκτός του ευρωατλαντικού χώρου για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δικών μας πολιτών εντός των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών οι σημερινές οικονομικές δυσκολίε μπορεί να είναι ένας πειρασμός για τις ευρωπαϊκές χώρες και να τις οδηγήσουν σε σωστρέφη. Αλλά χρειάζεται μια Ευρώπη έξω στρεφής, ε, με στένος και με ισχύ και αυτή η ανάγκη είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Γι' αυτό οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες με τρόπο επαρκή όσο και ευφυή και θα πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν προθυμία να χρησιμοποιούν αυτές τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουν όταν αυτό χρειάζεται. Τα καλά νέα είναι ότι η Ευρώπη δεν αρχίζει εδώ από μηδενική βάση. Σήμερα έχουμε μια Ευρώπη πιο ικανή και πιο πρόθυμη από ό,τι πριν από μια εικοσαετία είναι περισσότερα τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερους τόπους από ποτέ στην πρόσφατη ιστορία. Ακόμα και μικρές χώρες όπως η δική μου έχουν δώσει τη δυνατότητα ε, να, και έχουν αποδείξει μόνο τη δυνατότητα που έχουν να φανούν ενώτερες του μεγέθους τους. Και πρόσφατα στη Λιβύη οι ευρωπαϊκές χώρες απέδειξαν ότι είναι και πρόθυμες και ικανές να ηγηθούν σε μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, χωρίς τη σημαντική αμερικανή υποστήριξη, η επιχείρηση αυτή θα ήταν λιγότερο αποτελεσματική. Ο νεφοδιασμός η πτήση, η εποπτεία, η παρακολούθηση και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις έκαναν τη διαφορά. Για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να έχουν αυτή τη δυνατότητα, χρειάζεται πολιτική βούληση και πολιτική δέσμευση, όσο και οικονομική πόρη. Διότι τα κράτη από μόνα τους δεν μπορούν πλέον να επομίζονται αυτό το βάρος των στρατιωτικών δαπανών ε, είτε σήμερα είτε στο μέλλον. Αν όμως συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και τις μοιραζόμαστε, αν βοηθούμε ένα τον άλλον, αν έχουμε πολυεθνικές δυνάμεις και λύσεις, τότε μπορούμε να επομιστούμε αυτή την ευθύνη και τις ανάγκες που έχουμε για τον 21ο αιώνα. Αυτό λέγεται ευφυής άμυνα. Και σημαντικό στοιχείο της εφιούς άμυνας ε, είναι μεγαλύτερη συνεργασία και πιο στενή ε, συνεργασία και σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλληλοενισχυόμαστε αντί να αλληλοανταγωνιζόμαστε. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε 21 κοινά μέλη που έχουν τον ίδιο στρατό, τις ίδιες ενόπλες δυνάμεις και τους ίδιους φορολογούμενους όλες αυτές οι χώρες. Γι' αυτό καλωσορίζω την ε, πρωτοβουλία Pooling and Sharing της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνεκμετάλλευση και επιμερισμό στον αμυντικό τομέα. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα ε, από αεροσκάφους σε αεροσκάφους. Κυρίε και κύριοι, όλοι έχουμε να κερδίσουμε περισσότερα από μια ικανή ευρωπαϊκή άμυνα. Και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο οργανισμοί οφείλουν και μπορούν να παίξουν ένα ρόλο αλληλοσυμπληρούμενο και αλληλοβοηθούμενο για να ενισχυθεί η παγκόσμια ασφάλεια. Για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει επαρκώς στην κοινή μας ασφάλεια και θα πρέπει να συνεχίζει να επενδύει στους ζωτικούς δεσμούς που έχουμε ε, τους διατλαντικούς ε, και τους οικονομικούς και τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη και στη δέσμευση και προσήλωση της Ευρώπης για την προώθηση της ειρήνης ε, και της ασφάλειας και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και επέκεινα. Επίσης πιστεύω στην φιλοδοξία της Ευρώπης να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Υπάρχει πολύ υλικό προσυζήτηση. Φοβάμαι. Βλέπω ήδη τον κατάλογο των ομιλητών. Γι' αυτό το λέω. Και γι' αυτό θα επιβάλλω κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Γιατί αλλιώς θα τα καταφέρουμε. Πόσο να πούμε, δύο λεπτά. Συμφωνούμε. Κύριε Σαλαφράνκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Γενική Γραμματέα. Είναι πολύ ιδιαίτερη επικαιρότητα σήμερα εν ώψη και της επόμενης Συνόδου Κορυφής του Σικάγο. Και για το σκοπό αυτό συνεδριάσατε αρχές Απριλίου ε, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Βαρόσο και το εκφράσατε την επιθυμία σας, όπως επαναλάβατε και σήμερα, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας Ευρωπαϊκή Ένωση-ΝΑΤΟ θα ήθελα παρακαλώ, χωρίς υπερβολές, χωρίς να υπερτονίζετε τα θετικά, ούτε να κρύβετε τα αρνητικά, να μας ε, ε, πείτε μερικά λόγια, ε, καλύτερα τα διδάγματα από την επιχείρηση στη Λιβύη γενικότερα. Και κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η διαφορά στις απόψεις και στις αντιλήψεις και στη συμμετοχή των διαφόρων συμμάχων σε ό,τι αφορά ε, ε, τη γεωγραφική δράση από τη Λιβύη μέχρι το Αφγανιστάν ε, και άλλες πιθανές εμβάσεις του ΝΑΤΟ σε καταστάσεις τύπου Συρίας ή Σομαλίας. Ερώτηση τρίτη. Πώς βλέπετε τις σχέσεις με τη Ρωσία και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τι ρόλο διαδραματίζει αυτό τον καιρό ακόμα η Τουρκία για μεγαλύτερη ανάπτυξη των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό και ποιος είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον. Θα πρέπει να διατηρηθεί, θα πρέπει να πρωταγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του Βορειοατλαντικού Συμφώνου Ακούσαμε ε, όλη τις επικρίσεις του Υπουργού Εθνικής Αμήνης των ε, ίπα σε σχέση με την επιχείρηση στη Λιβύη και στο μέλλον τι θα γίνει με βάση την αρχή συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού. Και εν ώψη αυτού του τόσο σημαντικού ραντεβού που είναι η σύνδεση κορυφή στο Σικάγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κοπά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τα πυρηνικά όπλα στην ε, Ευρώπη. Ε, πόσο απαραίτητα είναι για το ΝΑΤΟ ε, η πυρηνική σταθμή στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί να αλλάξουν οι νατοϊκές δυνάμεις την επόμενη δεκαετία και τα σχέδια για την ε, πυραυλική άμυνα. Διερωτώ με αν η Συμμαχία θα πρέπει να πάρει άλλα μέτρα για να υπάρξουν αποτρεπτικά, αποτρεπτικοί παρά, παράγοντες, ούτως ώστε και να υπάρξει ασφάλεια, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των πυρηνικών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, οι απειρέ από το Ιράν ή την Βόρειο Κορέα, από τέτοια κράτη, τι ρόλο μπορούν να παίξουν σε αυτό το θέμα, το θέμα των πυράβλων. Ο κύριος από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα για τα σχόλιά του. Πριν από δύο μήνες συναντηθήκαμε στη Ουάσιγκτον. Εκεί μιλήσαμε το, για το πώς θα παρουσιάσουμε δημόσια την έννοια της α, έξυπνης άμυνας. Έχετε λάβει μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Και θα είναι πολύ σημαντικό και στη Σύνοδο Κορυφής του Σικάγο. Και το θέμα του στρατιωτικού δυναμικού. Είναι τέτοιο που δεν είναι εύληπτο από τον απλό άνθρωπο. Τι μέτρα λοιπόν έχετε λάβει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον, το δεύτερο εξάμεινο ε, του 2013 και όλο το 2014 είναι άγνωστο το τι θα συμβεί στο Αφγανιστάν. Η ΣΑΦ θα λειτουργεί αλλά η αποστολή θα μειωθεί για να υποστηρίζει τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν. Έχουν ληφθεί αποφάσεις ε, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής ε, στο Σικάγο προς αυτή την κατεύθυνση. Και τι θα γίνει μετά το 2014, μετά την αποστολή της ΙΣΑΦ. Θα υπάρξει μια συμμαχία. Τρίτον, Κύριε Γενικά Γραμματέα, γνωρίζετε την υποστήριξη που υπάρχει για τη μεταρρύθμισή σας. για τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το παρουσιάσετε δημόσια και να παρουσιάσετε και το επίπεδο της φιλοδοξίας που θέλετε να επιτύχετε στη Σύνοδο Κορυφή τη Λισαβόνα συμφωνήθηκε όμω ότι το στατιωτικό δυναμικό δεν θα μειωθεί μετά τη μεταρρύθμιση. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσετε δημόσια. Και σε ό,τι αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που προωθείτε στο ΝΑΤΟ. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας με τις σημερινές φιλοδοξίες του Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Αντίστοιχε ερωτήσει ε, με αυτέ ε, που ρώτησα στον ε, προκάτοχό σα πριν από έξι χρόνια. Κάνουμε μία έρευνα μετά από την έκθεση του Φεβρουαρίου του 2007 για συνενοχή στις μυστικές στήσεις της CIA. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τη θέση του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία στις 4 Οκτωβρίου του 2001 όταν ε, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε και το άρθρο 5 και κάποιες από τις επιφωνημένες δράσεις θα έπρεπε να ε, αυξήσουν τη συνεργασία ε, απέναντι στις απειλές της τρομοκρατίας. Και οι σύμμαχοι τον ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε εδάφη για ανεφοδιασμό κτλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ανησυχίε για το κατά πόσον το ΝΑΤΟ διμερός ή πολυμερός ε, διευκόλυνε αυτές τις παράνομε πτήσεις και τις παράνομες πρακτικές ε, συμπεριλαμβανομένων και των βαθανιστήριων. Και οι χώρες ε, όπως η Λιθουανία και η Ρουμανία ε, οι οποίες είχαν μυστικές φυλακές προσπάθησαν να ενταχθούν ε, ανάμεσα στο 2001 και 2004 στο ΝΑΤΟ τότε. Είχατε ποτέ την ευκαιρία να ερευνήσετε αυτές τους ισχυρισμούς ότι το ΝΑΤΟ ήταν μπλεγμένο με κάποιο τρόπο στη διευκόλυνση αυτής. Ε, δεν μιλάω για στρατιωτική συνεργασία, μιλάω για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών, υπηρεσιών πληροφοριών. Ερευνήθηκε το θέμα αυτό. Υπήρξε κάποια τέτοια έρευνα. Μπορείτε να μας ε, διαβεβαιώσετε κατηγορηματικά ότι το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν ήταν μπλεγμένο σε αυτό το θέμα και σε όλους τους ισχυρισμούς που έχουν ακουστεί για μυστικές φυλακές, για παράνομες πτήσεις, για μεταφορά ανθρώπων κτλ. Κυρία Λοχμπίλερ. Ε, νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να μιλήσει και για τη Σύνοδο Κορυφής του Σικάγου όμως. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Λάτφορντ, κάναμε μία ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από τα όσα αποκαλύφθηκαν για αυτό το πρόγραμμα της CIA και καλέσαμε τον ΝΑΤΟ. Είχατε σκεφτεί να συμμετάσχετε, αλλά τελικά αποφασίσατε να μην παραστείτε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω να απαντήσετε τουλάχιστον αυτές τις ερωτήσεις της συγκητριάς μας για το θέμα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Μπορείτε να σχολιάσετε το αποτέλεσμα της συνάντησης ε, του Συμβουλίου Ρωσίας-ΝΑΤΟ ε, την περασμένη εβδομάδα. Και μπορείτε να μας πείτε αν το νατοϊκό ε, αμυντικό σύστημα θα είναι ένα θέμα στη μερίσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής του Σικάγο. Κύριος Πιανέτα. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα είναι από την, ο κύριος είναι από την Ιταλική Βουλή. Μιλήσατε για τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρώπη σε μια προσπάθεια αμυντική. Πέρα από την κατανάλωση ασφάλειας, θα πρέπει να είναι και παραγωγός ασφάλειας, γενεσιουργός ασφάλειας. Όλοι μπορούν ε, να υποφεληθούν από μια πιο σίγουρη Ευρώπη. Μία ερώτηση, κύριε Γενική Γραμματέα. Τη δυνατότητα αυτής της συνεργασίας ε, στα πλαίσια της ε, συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού, ας πούμε, ε, στο Κωσυφοπέδιο και στα Βαλκάνια. Α, τι όλο μπορεί να παίξει. Και δεύτερον, υπάρχει κάποια ανησυχία λόγω του ότι στο Σικάγο δεν θα παραστεί η Ρωσία. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Υπάρχει ανησυχία από πλευράς ΝΑΤΟ λόγω της απουσίας της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Κλείνω τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Και δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Σαλαφράγκα, να σας απαντήσω καταρχάς σε εσάς. Από την επιχείρηση στη Λιβύη, τι μπορούμε να διδαχτούμε. Θέλω να τονίσω δύο σημαντικά διδάγματα. Καταρχάς, είναι δυνατό οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μαζί με τον Καναδά μάλιστα να παράσχουν τα περισσότερα στοιχεία, ε, τον εξοπλισμό σε μια σημαντική επιχείρηση και να έχουν το προβάδισμα. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο με την επιχείρηση στη Λιβύη, ότι παρά την ε, περίοδο οικονομικής λιτότητας η Ευρώπη ε, ανασκουμπόθηκε, έπαιξε το ρόλο της και πήρε Πολλέ ευθύνε στα πλαίσια αυτής τη επιχείρησης. Ε, το δεύτερο δίδαγμα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν έχουν κάποια ε, στρατιωτικά, κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό και στοιχεία. Εάν θέλει στο μέλλον η Ευρώπη να παίξει ρόλο στην ε, παγκόσμια διαχείριση της κρίσης, των κρίσεων γενικά, είναι να για να μπορέσει να το κάνει είναι να επενδύσει σε αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Παραδείγματο χάρη, α πούμε, στο ανεφοδιασμό σε καύσιμα εν, κατά τη διάρκεια τη πτήση. Υπάρχει μια τέτοια. Επίση η πρωτοβουλία μέσω του pooling and sharing, τη εκμετάλλευση και του επιμερισμού. Για να υπάρξουν αυτά τα, να δοθούν, να υπάρξουν στη διάθεση τη Ευρώπη αυτοί οι εξοπλισμοί. Έπειτα, ένα άλλο θέμα. Ε, αναγνώριση ε, πληροφορίες, ανεπάνδρωτα ελικόπτερα. Χρειάζεται τέτοια, τέτοιο εξοπλισμό η Ευρώπη. Ε, ενθαρρύνω τους Ευρωπαίους να επενδύσουν σε τέτοιο κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα βασικά διδάγματα που κρατάμε από την επιχείρηση στη Λιβύη. Με ρωτήσατε επίσης αν μπορούμε να φανταστούμε το ΝΑΤΟ να εμπλακεί σε νέες επιχειρήσεις αναφέρατε την ε, Συρία και, την, τη Συρία και τη Σομαλία. Καταρχάς για τη Σομαλία. Υπάρχει μια επιχείρηση της Αφρικανικής Ένωσης, υπό την αιγίδα μάλλον της Αφρικανικής Ένωσης και εμεί υποστηρίζουμε την Αφρικανική Ένωση και την επιχείρησή τη στη Σομαλία. Αλλά κατά προτεραιότητα είναι μια προσπάθεια αφρικανική και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Συρία. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση την πρόθεση να παρέμβουμε στη Συρία. Συχνά μου κάνουν την ερώτηση γιατί πήγατε στη Λιβύη και όχι στη Συρία. Η απάντηση είναι σαφής. Στη Λιβύη είχαμε μια εντολή του ΟΗΕ. Ενώ δεν έχουμε εντολή του ΟΗΕ για τη Συρία. Πέραν αυτού όμως, νομίζω ότι η Συρία είναι κάτι το τελείω διαφορετικό. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση και πολιτικά και θρησκευτικά και η εθνική σύνθεση της χώρας είναι τελείως διαφορετική και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι μια περιφερειακή λύση με έντονη συμμετοχή χωρών της περιοχής είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Λυπάμαι που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν κατάφερε να πετύχει τη συνένεση, ούτως ώστε να υπάρξει ένα ψήφισμα νομικά δεσμευτικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υποστήριξαν την δήλωση της Προεδρίας, που τώρα είναι η βάση για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και με βάση αυτό το σχέδιο πιστεύω να βρεθεί μια ειρηνική λύση στα προβλήματα της Συρίας. Καλό του Σύριους ηγέτες να λάβουν υπόψη τις θεμητές προσδοκίες του λαού τους και για δημοκρατία και ελευθερία και καταδικάζω την καταστολή του Συριακού λαού. Με ρωτήσατε για την ε, Τουρκία και τη σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωση δεν έχει φτάσει στο πλήρες δυναμικό της. Δεν νομίζω όμως ότι φταίει μόνο η Τουρκία γι' αυτό. Έχω υποβάλει κάποιες ρεαλιστικές λύσεις για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και μάλιστα, πρότεινα η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει ειδικέ ρυθμίσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και επομένως κάποιες ρυθμίσεις ως εκ τούτου για την ασφάλεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και από την άλλη η Τουρκία θα πρέπει να δεχτεί ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ γίνεται και με τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη, ρεαλιστική λύση, ένα πακέτο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει δυστυχώς καμία πρόοδος. Τέλος, με ρωτήσατε για το ρόλο των Αμερικανών μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τίποτα το καινοφανές ότι οι Ηνωμένε είναι η κυρίαρχη χώρα και σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν, υπάρχουν παρόλα αυτά εξελίξεις. Από το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρξαν εξελίξεις και προέκυψε ακόμα πιο σαφώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν τη μερίδα του λέοντος. Από το φορτίο ασφάλειας, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αν μου επιτρέπετε αυτή τη μεταφορά. Σήμερα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν μόνο το 20% των δαπανών ε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι πάρα πολύ το από μόνο του. Ο τρόπος για να προχωρήσουμε είναι οι Ευρωπαίοι να επενδύσουν σε σταδιωτικό δυναμικό και σε μια περίοδο οικονομικής λιτότητας ο μόνος τρόπος για να το πετύχουν είναι ε, μέσω της πολυεθνικής ε, συνεργασίας. Ε, μέσω δηλαδή αυτής της έξυπνης προσπάθειας του pooling and sharing, της συνεκμετάλλευσης και του επιμερισμού. Για την πυραυλική άμυνα, με ρώτησε η κυρία Κοπά. Η πυραυλική άμυνα δεν είναι ε, κατά μια οποιασδήποτε χώρα, αλλά κατά μια οποιασδήποτε απειλής από όπου και αν προέρχεται. Το γεγονός ότι περισσότερο από 30 χώρες στον κόσμο έχουν πυραυλική τεχνολογία ή προσδοκούν και ελπίζουν να αποκτήσουν τέτοια τεχνολογία και ορισμένες έχουν και την δυνατότητα να πλήξουν ε, νατοϊκά εδάφη, Ακριβώς γι' αυτό χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ε, μία ανατοϊκή πυραυλική άμυνα, ένα τέτοιο ανατοϊκό σύστημα, το οποίο δεν κατευθύνεται εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά οποιασδήποτε απειλής. Με ρώτησατε επίσης άλλοι τι βήματα έχουμε πάρει για να προωθήσουμε την έξυπνη άμυνα. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο που θα πρέπει να υιοθετηθεί στις κορυφή του Σικάγου τον επόμενο μήνα. Σε αυτό το πακέτο θα έχουμε πάνω από 20, πάνω, 20 ε, ε, συγκεκριμένα πολυεθνικά προγράμματα. Τους τελευταίους μήνες βρήκαμε τα κράτη τα οποία θα αναλάβουν τα project αυτά, τα προγράμματα αυτά. Έχουμε βρει τους συμμετέχοντες σε αυτά τα πολυεθνικά προγράμματα και θα καλύπτουν τομείς πολλούς, ευρύς, όπου χρειαζόμαστε καλύτερο δυναμικό, ε, κοινή επιμελητία, ε, κατάρτιση, αναβάθμιση στρατιωτικού εξοπλισμού. Όλα αυτά θα γίνουν χάρη στις κοινέ μας προσπάθειες. Υπό αυτή την προσπάθεια του Smart Defense, της έξυπνης άμυνας, στο Αφγανιστάν. Μετά το 2014, η αποστολή τι ρόλο θα έχει. Υπάρχει μια συμφωνία θέλουμε να συνεχίσουμε μία ε, αποστολή κατάρτισης υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Μέχρι το τέλος του 2014 θα σταματήσει η αποστολή της ΣΥΣΑΦ. Αλλά θα παραμείνουμε ε, δεσμευμένοι και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει με αυτή την αποστολή ε, κατάρτισης μετά το 2014. Ακόμα συζητάμε βέβαια τους τρόπους, αλλά είναι σαφές ότι θα είναι μία αποστολή κατάρτισης προς υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας. Επομένως, δεν θα είναι μια συμμαχία εθελοντών, αλλά θα είναι μια τέτοια αποστολή υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Το συζητάμε αν χρειαζόμαστε περισσότερο δυναμικό για να προστατεύσουμε τους εκπαιδευτές μας και να βοηθήσουμε τις αυγανικές ε, δυνάμεις ασφαλείας. Θα πάρουμε την απόφαση της συνοκορυφή του Σικάγου. Για τη μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ. η φιλοδοξία μας δεν έχει αλλάξει. Δεν αλλάζει το επίπεδο. Το επίπεδο φιλοδοξίας παραμένει το ίδιο. Θα κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τόσο ώστε οι δομές μας να είναι πιο αποτελεσματικές, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας και στο μέλλον. Η Λέδη Λάτφορντ με ρώτησε για την ενεργοποίηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου του 2001. Μία μέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που κάναμε, εξακολουθούμε να το κάνουμε καταρχήν. Τι κάνουμε; Αναπτύξαμε δημιουργήσαμε μία επιχείρηση αντιτρομοκρατική, θαλάσσια, στο Denver, η οποία, συγγνώμη, ε, είναι ακόμα ενεργή στην Μεσόγειο. Και σας διαβεβαιώ ότι το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν έχει εμπλακεί ή δεν είναι εμπλεγμένο σε παράνομες δραστηριότητες. Κυρία Λοχμπίλερ, με ρώτησε για την σύνοδο που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Ε, Κάνω μια αποτίμηση της ε, συνεργασίας ε, ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ε, Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια υπήρξε σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ενισχύσαμε τη συνεργασία για το Αφγανιστάν. Οι Ρώσοι μάλιστα μας βοήθησαν με κάποιες ρυθμίσεις διαμετακόμισης και διέλευσης. Επίσης, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις κατά της πειρατείας, κατά των ναρκωτικών κτλ. Γενικά έχει ενισχυθεί η συνεργασία μας με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια όπου δεν συμφωνούμε με τη Ρωσία. Το θέμα της Γεωργίας. Θέλουμε να υπάρξει πλήρης σεβασμός ε, η, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της ε, γεωργία. Η πυραυλική άμυνα είναι άλλο θέμα που διαφωνούμε. Έχουμε καλέσει τη Ρωσία να συνεργαστεί, αλλά δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο στις σημειώσεις μας ή συζητήσεις όμως για την πυραυλική άμυνα θα συνεχιστούν και ελπίζω κάποια στιγμή να συναυθεί μια συμφωνία για να υπάρξει συνεργασία για την πυραυλική άμυνα. Γενικά ήταν καλή αυτή η συνάντηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Ε, Κύριε Πιανέτα, με ρωτήσατε για την εφαρμογή της ε, έξυπνης άμυνας και για το pooling και sharing σε σχέση με το κοσφοπέδιο και τα Βαλκάνια εν γέννη. Ας διευρύνω λίγο το πλαίσιο και ας μιλήσω για την ανάγκη εργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοσμοπέδιο. Να σας πω ειλικρινά. Η... Πρέπει να σας πω ότι η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης EULEX δεν έχει αρκετούς πόρους Αυτό έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις και για το ΝΑΤΟ, γιατί η δική μας επιχείρηση K4 πηρεάζεται αναγκαστικά. Αναλαμβάνουμε ευθύνε και καθήκοντα που δεν είχαν προβλεφθεί. Ειδικά στο βόρειο τμήμα του κοσφοπεδίου. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε στενό συντονισμό, ούτω ώστε να υπάρχει ε, ο σωστός καταμερισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε έναν ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας ισχυρής EU-LEX, ώστε να υπάρξει να υπάρξει καλύτερο καταμερισμό, όπω σα είπα, αρμοδιοτήτων. Ελπίζω να ασκήσετε και εσεί την πίεση, ούτω ώστε να επανδροθεί όπω πρέπει η EULEX. Ε, για τη Ρωσία και το Σικάγο. Δεν θα έχουμε μία σύνοδο κορυφή ΝΑΤΟ-Ρωσία. Ε, μίλησα με τον εκλεγμένο πρόεδρο Πούτιν πριν λίγε εβδομάδε και συμφωνήσαμε ότι λόγω του ότι των πολλαπλών υποχρεώσεών του εντό τη Ρωσία, ε, θα αναλάβει την, ε, το αξίωμά του ο Σονούπο και θα το έχει αναλάβει λίγες εβδομάδες πριν από τη συνοκορυφή του Σικάγο, ε, δημιουργεί προβλήματα στο να δημιουργηθεί, στο να γίνει μια συνοσκορυφή ΝΑΤΟ-Ρωσία στο Σικάγο. Αλλά συμφωνήσαμε διμερώ να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατόν. Και θα έχουμε, είχαμε και μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα που σα είπα ΝΑΤΟ-Ρωσία. Επομένω, η συνεργασία μα με τη Ρωσία θα συνεχιστεί. Η σχέση μας με τη Ρωσία δεν εξαρτάται από μία συνάντηση, ακόμα και αν είναι μία σύμβαση κορυφή. Καλέσαμε τη Ρωσία ούτω ώστε να, ε, να συμμετάσχει στη συνάντηση ΙΣΑΦ στο Σικάγο. Ε, με όλα αυτά βλέπετε ότι θα συνεχίσουμε το διάλογό μας με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Oh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε και από την ομάδα ECR. Είμαστε νομίζω οι πλέον φερμοί υποστηρικτέ του ΝΑΤΟ. Για τη Λιβύη, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι οι, αερο, οι αεροπορικέ δυνάμει δεν, ήταν δεν οι μόνε που μπόρεσαν να α, χτυπήσουν του στόχου. Χρειάστηκαν και ειδικέ δυνάμει από τι υπόλοιπε χώρε. Ε, συμφωνείτε με αυτό, και μήπω ε, υπάρχει τελικά κίνδυνος ε, διάδοσης όλων αυτών των όπλων. Μπορεί βεβαίως να είναι μικρά όπλα, αλλά μπορεί όντω να υπάρχουν συνδεσμοί με κάποιες ε, παρακλάδια της Αλκάιντα. Στη σύνοδο της, του Σικάγο διάβασα στους Financial Times σήμερα ότι η Αμερική συμφώνησε για το 2014, αλλά μήπως το Αφγανιστάν γίνει μια, ένα, μια ας πούμε δυτική ε, και μήπως δεν πρέπει να ε, επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας και να κάνουμε τελικά όλη την ε, δύσκολη δουλειά που χρειάζεται να δημιουργήσουμε δηλαδή ασφάλεια στη χώρα. Το 2014 το μεγάλο όγκο των ε, δυνάμεων θα έχει φύγει. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες δυνάμεις γύρω-γύρω, Ρωσία, Ινδία, Πακιστάν, θεωρείται θα αλλάξει δυναμική μόλις α, ολοκληρωθεί και η εντολή της ISAF και επίσης για την, ε, ε, για την επικάλυψη δυνάμεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του ΝΑΤΟ. Και οι δύο προσπαθούν να επενδύσουν περισσότερο στην κλιματική ασφάλεια, στι στις κλιματικές αλλαγές, στην ασφάλεια του επιστημισμού κτλ. Στα πιο ελαφρά δηλαδή ε, ζητήματα. Αλλά μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση και, την, και τις περικοπές που γίνεται σε δημοσιονομικό επίπεδο, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους επικαλύψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάριος Βόλσκι, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. καλώ ήρθατε. Καταρχάς, σε χαρητήρια για το ότι έχετε καταστήσει το ΝΑΤΟ έτσι πιο εύληπτο σε όλους μας και πιο κοντά μας το έχετε φέρει. Η πραγματικότητα δεν είναι προφανώς ε, η καλύτερη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε ακριβώς να κατανοούμε σωστά τα καθήκοντα μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΤΟ. Όπως ξέρετε η Ευρώπη βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση. Αυτό προφανώς μειώνει τους αμυντικούς υπολογισμούς και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ποια είναι η λύση που θα δίνατε εσείς ε, έτσι ώστε να μπορούμε και μακροπρόθεσμα να διατηρήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ο ε, επικεφαλής της ε, Λιθουανικής αντιπροσωπεία στο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Dear Secretary General, dear Mr. Brock. Κύριε Γενική Γραμματεία, κύριε Μπροκ. Εμείς είμαστε ε, γείτονες με την περιφέρεια του Καλίνιγκρατ και έχουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τεράστιες εξελίξεις στην, ε, ε, σε αυτή την, ε, στην ύπαρξη όπλων στην, σε αυτή την πολύ μικρή περιοχή στην, μέσα στο ΝΑΤΟ. Άκουσα βεβαίως την εισαγωγική σας παρέμβαση για, το, για την σύνοδο με τη Ρωσία. Η συνεργασία αυτή βεβαίως είναι καλή. Αναφέρατε τα ναρκωτικά, αναφέρατε άλλα μέτρα αναφέρατε την μεταφορά στο, στις μεταφορές στο Αφγανιστάν, αλλά για την ασφάλεια των εσωτερικών μας υποθέσεων ε, και για το ΝΑΤΟ και για να μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε τα κοινά μας σύνορα, ε, τι θα πρέπει να γίνει. Εμάς μας ανησυχούν λίγο αυτές οι νέες εξελίξεις, οι νέοι πύραυλοι στο, στο Καλίνιγκραντ, Πρόσφατα είδαμε μάλιστα τέτοιες νέες εξελίξεις, οπότε θα ήθελα να θέσω το ερώτημα τι γίνεται με την περιοχή του Καλίνιγκρατ και πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την τελευταία πρόσφατη εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ. Θα ήθελα μία ε, διευκρίνηση για την ε, πυραυλική άμυνα. Ε, το 2010 μιλήσατε για επιπλέον κόστος για μια ε, πυραυλική άμυνα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, ε, εσωτερικές μελέτες του ΝΑΤΟ λένε ότι αυτά τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Οπότε ποιο είναι το ποσό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα. Και επίσης για την πολιτική των πυρηνικών. Ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα που περιμένουμε από την στρατηγική για τα πυρηνικά ειδικά σε ό,τι αφορά τα, τα πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη. Η δική σας θέση ποια είναι. Εσείς ε, είσαστε υπέρ της απόσυρσής τους. Και ένα ερώτημα να συμπληρώσω για τα ερωτήματα που υπόθηκαν ήδη για το Αφγανιστάν. Μιλήσατε για μια εκπαιδευτική ε, επιχείρηση. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια μιας ε, γενικότερης επιχείρησης του ΝΑΤΟ και κατάλαβα καλά ότι σε αυτή την ε, εκπαιδευτική ε, επιχείρηση θα παραμείνουμε μόνο στα εκπαιδευτικά θέματα. Δηλαδή δεν θα υπάρξουν ε, ή θα υπάρξουν επιπλέον επεμβάσεις. Και επίσης, η αποστολή στο Αφγανιστάν στα πλαίσια ποιας ομάδας του ΝΑΤΟ θα, από ποια, στα πλαίσια ποιας ομάδας του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μιλήσατε όλοι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί ομιλητέ ακόμη, οπότε να συμφωνήσουμε ότι θα δώσουμε 1,5 λεπτό στον καθέναν από εδώ την προς για να προλάβουμε όλου. Ο κύριο Λίζεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, ως Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα, θα ήθελα να πω ότι αυτό που λέγατε είναι πραγματικά ζωτική σημασία για την δική μας την υποεπιτροπή. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ε, κοινή ε, πολιτικής άμυνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των τελευταίων μηνών που προκύπτει από την Υποεπιτροπή Άμυνα και Εθνή πόσο σημαντικό θέμα είναι αυτό για μας. Γι' αυτό πραγματικά εκτιμώ αυτά που είπατε μέχρι στιγμής και βεβαίω καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ έχει βελτιωθεί. Είτε είναι αυτό στο Αφγανιστάν, είτε στη Σομαλία, είτε οπουδήποτε η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ συμμετέχουν και δρούν από κοινού. Έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα στο παρελθόν, η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί. Έχω ένα ερώτημα για τη Γεωργία. Το θέμα της Γεωργίας θα α, θυγεί στο, στην Σύνοδο του Σικάγο. Η Γεωργία είναι μια χώρα για την οποία έχουμε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα μας ήδη από το Βουκουρέστι. Η κατάσταση στον Κάφκασο παραμένει περίπλοκη, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το θέμα της Γεωργίας θα το συζητήσετε στο Σύνοδο του Σικάγο και αν ναι με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντρόμπα, ε, αντιπρόεδρος της ε, Σλοβακικής Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το δυστύχημα της, του σκάφου στην Μεσόγειο τα, στα τέλη Μαρτίου. Ξέρω βέβαια ότι δεν είναι το ΝΑΤΟ ο κύριος ύποπτος εδώ, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς έχει γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση τέτοιων πιθανότητων στο μέλλον. Οπότε, ερώτημα, το ΝΑΤΟ τι μπορεί να κάνει για να αποφύγει, να αποτρέψει τέτοια ατυχήματα στο μέλλον και αν θα υπάρξει κάποια δήλωση ίσως από πλευράς του ΝΑΤΟ. Ε, Ο κύριος Κυρίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα, ευχαριστώ που είστε εδώ και για τις καθαρές απαντήσεις που μας δίνετε. Συμφωνώ με την ε, δική σας αξιολόγηση για το ότι θα πρέπει όντως να υπάρξει ε, όραμα από πλευράς ευρωπαϊκής για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων. Έχω όμως ένα ερώτημα. Έχοντα υπόψη ότι υπάρχει σαφής ε, τάση ε, του να αλλάξει το στρατιωτικό ενδιαφέρον και να πάει προς την Ασία και από πλευράς ε, εξοπλισμού και δυνατοτήτων. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φανεί ότι δεν είναι επικεφαλής πια. Μιλάτε για ένα πακέτο το οποίο θα υιοθετηθεί στην Σύνοδο του Σικάγο. Αλλά Πέραν του ότι αυτό μπορεί όντω να γίνει, μπορεί να υπάρξει όντω η ε, συνεκμετάλλευση των ε, ε, πηγών, των πόρων κτλ. Η δική σα αξιολόγηση ποια είναι, προφανώ δεν μπορείτε να μα πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο χρονικά, αλλά στο μέλλον πότε θεωρείτε ότι ω δυνατότητα θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσατε να αναλάβετε μια τέτοια επιχείρηση τέτοιου μεγέθου. Ο κύριο Νταφ έχει το λόγο. Η μεγαλύτερη στρατιωτική απειλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα νομίζω ότι προέρχεται από τις εξελίξεις που παρακολουθούμε στο Ιράν. Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο να ζητήσουμε από το Ισραήλ να είναι παρόν στη σύνοδο του Σικάγο για να συζητηθεί το θέμα αυτό, γιατί η κατάσταση πραγματικά επιδεινώνεται τραγικά στο Ιράν. Και είναι αλήθεια ότι η Τουρκία έχει μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση πρόσκλησης προς το Ισραήλ. Και για την Τουρκία κάτι ακόμη. Ο αντίκτυπος ποιος είναι στην ε, αξιοπιστία που υπάρχει από πλευράς Τουρκίας ως εταίρου του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την σύλληψη και την φυλάκιση πολλών από τους στρατηγούς, από το στρατιωτικό επιτελείο της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα η κυρία Λέζινγκ το ανέφερε, αλλά το κόστος με ενδιαφέρει και εμένα, το κόστος για την πυραυλική άμυνα. Και επίσης, να δούμε ποια θα είναι η επικράτεια που θα καλύπτεται. ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκά κράτη ή θα υπάρχει κάποια περιφέρεια που δεν θα καλύπτεται. Και ένα δεύτερο ερώτημα για το σκάφος με τους μετανάστες. Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μια εσωτερική έρευνα Υπάρχει κάποια διαδικασία διερεύνησης ε, αυτού του ατυχήματος και αν ναι θα μας θα ανακοινώσετε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Ευχαριστώ. Yeah, um, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πρέπει να απαντήσω πολύ σύντομα γιατί είναι μεγάλη χρονική περιορισμή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Ο κύριος Τάνοκ πρώτα. Ανησυχείτε για το Αφγανιστάν. Μήπως ε, γίνει ένα ε, κράτος ε, πελάτης της δύση, έτσι το χαρακτηρίσατε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Προφανώς το Αφγανιστάν θα χρειαστεί τη βοήθειά μας. Και πέρα του 2014. Αναφερθήκατε σε μια έκθεση, ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει, πιστεύω, με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αφγανιστάν για μια ε, πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, εταιρική σχέση, διμερής είναι αυτή, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αφγανιστάν. Προσωπικά πιστεύω ότι μια τέτοια μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση θα στείλει ένα μήνυμα κρίσιμο αλλά και καθηγαστικό και προς τους Αφγανούς πολίτες αλλά και προς τους γείτονες του Αφγανιστάν. Επίσης θα στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τους εχθρούς του Αφγανιστάν ότι δεν, δεν μπορούν να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουν να φύγουν τα διεθνή στρατεύματα από το Αφγανιστάν και μετά να είναι ελεύθεροι. Θα παραμείνουμε με έναν τρόπο υποστηρικτικό. Οι ε, δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός του Αφγανιστάν θα αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό όμως δεν καθιστά τη χώρα ε, κράτος πελάτη της Δύσης. Από την 1η Πρώτου του 2015 οι ε, δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια στην επικράτειά τους. Εμείς θα είμαστε παρόντες για να τους υποστηρίζουμε, αλλά την πλήρη ευθύνη θα την έχουν εκείνοι. Έτσι ορίζεται το κυρίαρχο κράτος και το κράτος που αναλαμβάνει τις ευθύνες για την ίδια του την ασφάλεια. Και επίσης πιστεύω ότι αυτό θα έχει και θετικό αντίκτυπο στην όλη δυναμική στην περιοχή, διότι η γείτονε του Αφγανιστάν και ιδιαίτερα το Πακιστάν ανησυχούν βεβαίως πάρα πολύ για τις μελλοντικέ εξελίξεις στη χώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβεβαιώσουμε τους γείτονες ότι δεν θα φύγουμε και θα αφήσουμε πίσω μας ένα κενό ασφαλείας. Ούτε θα είναι αποτυχημένο κράτος το Αφγανιστάν. Αλλά θα είναι ένα κράτος που θα λειτουργεί σχετικά καλά και θα είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες της ίδιας της ασφάλειας χάρη σε μια πάρα πολύ ικανή ε, στελέχωση των δυνάμεων ασφαλείας. Βεβαίως και είναι πρόκληση, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Πρόσφατα είδαμε στην Καμπούλ εντυπωσιακέ επιθέσει, αλλά αυτό που επίση είδαμε ήταν πάρα πολύ ικανέ δυνάμει ασφαλείας που αντιμετώπισαν αυτέ τι προκλήσει για την ασφάλεια. Ε, με ένα πάρα πολύ επαγγελματικό τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι καλά νέα και είμαι πραγματικά ε, αισιόδοξο ότι θα μπορέσουν να χειριστούν αυτά τα θέματα ασφαλείας όταν η επιχείρηση ISAF ολοκληρώσει τις εργασίες της ε, στα τέλη του 2014. Διότι θα είμαστε παρόντες ακόμα για να τους υποστηρίσουμε. Και επίσης η διεθνής κοινότητα έχει δεσμευτεί να συμμετέχει και στη χρηματοδότηση των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και μετά το 2014. Όταν τερματιστεί η επιχείρηση ISAF στα τέλη του 2014, ε, οι δυνάμεις ασφαλείας θα αριθμούν ένα προσωπικό 350.000. Δηλαδή αυτό είναι ένα μέγεθος και οικονομικό μέγεθος που υπερβαίνει κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες της αφγανικής κυβέρνησης. Η Εθνική κοινότητα δεσμεύθηκε στη διάσκεψη της Βόνης να συμμετάσχει και ε, στη χρηματοδότηση των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και μετά το 2014. Με αυτή λοιπόν την υποστήριξη και τη δέσμευση ε, είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσει το Αφγανιστάν να σταθεί στα πόδια του αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα σταθεί μόνο του στα πόδια του. Τώρα, για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την ΕΠΑ, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, συμφωνώ πολύτως ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και τους ανταγωνισμούς. Θα πρέπει να βοηθούμε ένα τον άλλον και να βεβαιωθούμε ότι αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμπληρωματικά προς τα όσα κάνει το ΝΑΤΟ και τούμπαλιν. Ε, αυτή θα πρέπει να είναι η φόρμουλα. Πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, ότι στην κατεύθυνση αυτή ε, τα πηγαίνουμε πολύ καλά, ε, αρκετά καλά. Πέρα από τις γενικές πολιτικές προκλήσεις και την εταιρική σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε γενικές γραμμές έχουμε εξασφαλίσει Σε επίπεδο υπηρεσιών στελεχών έχουμε πολύ καλή συνεργασία και συντονισμό στα πλαίσια του πολιτικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί. Συγκεκριμένα, όταν έχουμε την πρωτοβουλία για την ευφυή άμυνα, του ΝΑΤΟ και την άλλη την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Pooling and Sharing, την ε, συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό, έχουμε πολύ καλό συντονισμό, εξαιρετική συνεργασία που εξασφαλίζει αυτή τη συμπληρωματικότητα στη δράση μας. Ο κύριος Άρους Βόλσκι με ρώτησε ε, στο ίδιο πνεύμα. Πώς να φανταστώ τον επιμερισμό εργασίας ή τον καταμερισμό των ευθυνών και καθηκόντων μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ανέφερα ήδη ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που ήταν η δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα από αεροσκαφο σε αεροσκάφο. Γιατί εμεί γενικά δεν έχουμε έλλειμμα στι δυνατοτητε των ΝΑΤΟ σε αυτή τη ε, δράση, γιατί οι Αμερικανοί έχουν πάρα πολλά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν οι Ευρωπαίοι. Οπότε γιατί να επικαλυπτόμεθα. Βεβαίως είναι αμυγός ευρωπαϊκή ευθύνη και καθήκον του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού και εμείς εκτιμούμε αυτή την προσπάθεια και την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά γενικότερα επιχειρούμε ε, στα ίδια ε, μέρη. Στο Αφγανιστάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αστυνομική ε, αποστολή, εμείς έχουμε στρατιωτική. Στο Κόσοβο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αποστολή κράτους δικαίου και αστυνομική. Εμείς έχουμε στρατιωτική αποστολή. Ιδού τα παραδείγματα καταμερισμού ευθυνών και εργασίας στην ίδια γεωγραφική περιοχή και στο ίδιο θέατρο επιχειρήσεων. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αφρική θα ήταν ένα σημείο που θα την ενδιαφέρει περισσότερο από ότι το ΝΑΤΟ, ας πούμε. Σε τέτοια θέματα γεωγραφικά, ειδικά, ειδικών αποστολών ή ρόλο που έχει ο καθένας να παίξει, εκεί βλέπω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε ε, τα καθήκοντα και να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Επίσης με ρωτήσατε για τις συνέπειες ε, των μειούμενων προϋπολογισμών. Νομίζω ότι αναφέρθηκα προηγουμένως αυτό. Πιστεύω ότι η σωστή απάντηση είναι οι πολυεθνικές λύσεις και όχι αμυγός εθνικές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι σύμμαχοι, ο καθένας από μόνος του, δεν θα είναι σε θέση να επομιστεί, δεν το αντέχει ο προπολογισμό να αγοράζουν ακριβούς εξοπλισμούς στο μέλλον. Μπορούμε όμως να το κάνουμε μαζί, να βοηθούμε ένας τον άλλον με κοινά σχέδια. Πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα μεταγωγικά αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε την πρωτοβουλία για το C17. Δέκα μεγάλοι σύμμαχοι και δύο εταίροι, η Σουηδία και η Φιλανδία όπως γνωρίζετε δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά δέκα σύμμαχοι και δύο εταίροι ε, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αγοράσουν τρία μεταγωγικά ε, C17. Δεν μπορούσαν κάθε χώρα ξεχωριστά να το αγοράσουν. Τώρα έχουν ένα κοινό στόλο τριών αεροσκαφών και μπορούν ε, να αγοράζουν ώρες πτήσεων σε αυτά τα αεροπλάνα. Ιδού ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφιούς άμυνας. Και αυτό το ε, θέμα, το πλαίσιο και η αντίληψη μπορεί να διευρυθεί και αλλού για να τετραγωνιστεί, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτός ο κύκλος. Για τον κύριο Ζιγκέρης και το Καλίνιγκρατ και την ε, παρουσία εκεί. Πραγματικά είναι ανησυχητική αυτή ετέθη ε, στη συνάντηση του Συμβουλίου με τη Ρωσία, γιατί ξέρετε συζητούμε ειλικρινά όλα αυτά τα θέματα και θα πρέπει να σας πω ότι είναι απόλυτη σπατάλη χρημάτων. Αν αποφασίσουν οι Ρώσοι να αναπτύξουν εκεί επιθετικές ε, δυνάμεις που να στρέφονται κατά κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία ε, πρόθεση, μα καμία, να επιτεθεί στη Ρωσία. Οπότε σπαταλούν τα χρήματά τους αν θέλουν να επενδύσουν δεν ξέρω πόσα λεφτά εκεί πέρα σε μια τέτοια ε, επιθετική παρουσία απέναντι σε έναν τεχνητό εχθρό, έναν φανταστικό εχθρό που δεν υπάρχει. Αυτά τα χρήματα θα τα δαπανούσαν καλύτερα ε, στην ε, κοινωνική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της ρωσικής κοινωνίας. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο για αυτό το θέμα. με την κυρία Δεν έχω καινούργια στοιχεία. Παραμένουν οι ίδιοι αριθμοί και τα ποσά. Το επιπλέον κόστος για να συνδεθούν ε, αντιπυραυλικά συστήματα που ήδη υπάρχουν και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που μπορεί να προστατεύει ως ασπίδα όλους τους πληθυσμούς των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και να καλύπτει όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια των ε, συμμάχων. Αυτό το επιπλέον κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Καινούριο νούμερο δεν έχω. Πρέπει να σας πω ότι αυτό ισχύει. Βεβαίως δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση, διότι πριν από πολύ καιρό οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να επενδύσουν σε εκείνο που ονομάζουμε αντιπυραυλικό σύστημα στα θέατρα των επιχειρήσεων, δηλαδή εκεί που έχουμε αναπτυγμένα στρατεύματα. Πριν από πάρα πολύ καιρό έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση και το κόστος θα είναι περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπλέον, μόνο για 200 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να διευρύνουμε την προστασία των ε, στρατευμάτων και ταυτόχρονα και όλου του πληθυσμού. Αυτό το λέω πολύ συμφέρουσα υπόθεση. Με ρωτήσατε για τα πυρηνικά στη συνέχεια. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μειωθούν ε, ε, τα τακτικά πυρηνικά όπλα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά τον αριθμό των ρωσικών τακτικών πυρηνικών ε, όπλων, διότι εκεί υπάρχει μεγάλη απόσταση. Η Νατοϊκή Σύμμαχη έχει μειώσει σημαντικά τα πυρηνικά τους από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά, αλλά δεν έχει συμβεί το ίδιο και στη Ρωσία. <laughs> δηλαδή υπάρχει αυτή η δυσαναλογία όντως και αν θέλουμε να μειώσουμε ε, τα πυρηνικά μας, που βεβαίως θα ήταν θαυμάσια ε, είδηση, θα πρέπει να γίνει με τρόπο εξορροπημένο Αυτή είναι η απάντησή μου για τα πυρηνικά. Για το Αφγανιστάν τώρα, η εκπαιδευτική αποστολή είναι εκπαιδευτική, αλλά οι εκπαιδευτέ μα θα πρέπει κάπου και να προστατεύονται. Και τώρα ε, συζητούμε αυτό τον καιρό για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό. Αφελεί δεν είμαστε. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν τους Αφγανού σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Ο κύριος Λίνσεκ με ρώτησε για τη Γεωργία. Νομίζω θα στείλουμε ένα μήνυμα πολύ ενθαρρυντικό από το Σικάγο στη Γεωργία, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η σύνοδο κορυφή του Σικάγο δεν είναι σύνοδο διεύρυνση. Δεν θα, δεν θα απευθύνουμε νέε προσκλήσεις ούτε στη ε, Γεωργία ούτε σε κανέναν άλλον υποψήφιο. Ε, ε, αλλά η Γεωργία έχει κάνει πολλά για τις μεταρρυθμίσεις και βεβαίως αυτό θα αντανακλάται και στη δήλωση, τη διακήρυξη του Σικάγου. Ο κύριος Ντρόμπα με ρώτησε για το επεισόδιο αυτό με το σκάφος με τους μετανάστες. Και η κυρία Μπραντνερ αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ ατυχές, όσο και τραγικό συμβάν. Αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Οι σύμμαχοι, τα μέλη του ΝΑΤΟ, έκαναν πολλά για να σώσουν ζωές κατά τη διάρκεια της επιχείρησή μας στη Λιβύη. Και μάλιστα προλάβαμε τη σφαγή επί του λιβυκού πληθυσμού. Και στη θάλασσα. Κάναμε πολλά για να σώσουμε κόσμο. Συμμαχικά πλοία συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης περίπου 600 ανθρώπων. Και θα ήθελα να το γνωρίζετε αυτό. Αυτή είναι πραγματικά η ουσία της επιχείρησής μας στη Λιβύη. Ζωές σώσαμε. Επίσης κάναμε πολλά ε, για να ε, δώσουμε πληροφορίες και ενημέρωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης που διερευνά αυτό το συμβάν. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε πάντα πρόθυμοι και ακόμα να δώσουμε και νέα στοιχεία όσα έχουμε στη διάθεσή μας, άμα μας τα ζητήσουν. Αυτή ήταν η απάντησή μου στην κυρία Μπράτνο. Ο κύριος Ντρόμπα με ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αποφεύγουμε τέτοια επεισόδια στο μέλλον. Μα δεν νομίζω ότι είναι πρωταρχικά υπόθεση του ΝΑΤΟ αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθούμε όσους κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά όχι μόνο εμείς. Αυτή είναι καθολική παγκόσμια ευθύνη και υποχρέωση όλων, δεν είναι ειδική ευθύνη του ΝΑΤΟ. Βεβαίως τα συμμαχικά πλοία που πλέον στην περιοχή βεβαίως θα πρέπει να αναλαμβάνουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, στο πέλαγος όπως και ε, κάθε άλλο σκάφος. Οι, όλες οι ναυτικές μονάδες το κάνουν αυτό. Ο κύριος Κύριλοφ με ρώτησε για το νέο στρατηγικό δόγμα και αμυντικό δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που δείχνει ότι προσανατολίζονται πιο πολύ προς την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Και με ρωτήσετε και η Ευρώπη θα φεθεί στη μοίρα της να ε, ε, διαχειρίζεται διεθνώς τις κρίσεις με επιχειρήσεις τύπου Λιβύη στο μέλλον. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι είναι φυσικό οι Ηνωμένε Πολιτείε να εστιάζουν τώρα την προσοχή τους περισσότερο στην Ασία και στον Ειρηνικό και τις αναδυόμενες εκεί δυνάμεις. Αυτό είναι και προς το συμφέρον της Ευρώπης ε, παρόδο. Αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο τμήμα της αμυντικής στρατηγικής ε, των ΗΠΑ. Είναι προσιλωμένη στην Διατλαντική Συμμαχία. Μπορεί οι Ηνωμένε να μειώσουν ε, τις δυνάμεις τους, τα, τα, τις που σταθμεύουν στην Ευρώπη, αλλά σε αντάλλαγμα θα ε, επενδύσουν στην αντιπυραυλική ασπίδα μονάδες για την ε, απόκριση του ΝΑΤΟ και σε κοινέ ασκήσεις και γυμνάσια στην Ευρώπη. Δηλαδή ε, θα παραμείνει ισχυρή η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και στο μέλλον όπως στο παρελθόν, αλλά οι καιροί αλλάζουν και όλοι θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις και προκλήσεις ασφαλείας. Για τον κύριο Νταφ. Με ρώτησε αν σκεφτήκαμε να καλέσουμε το Ισραήλ στο Σικάγο. Όχι. Δεν μας πέρασε από το μυαλό. Και επίσης για τον ίδιο λόγο μπορώ να σας απαντήσω σαφώς ότι ούτε μπλόκαρε η Τουρκία ούτε τίποτα τέτοια πρόσκληση γιατί ε, απλώς δεν μας απασχόλησε αυτό. Δεν σκεφτήκαμε καν να καλέσουμε το Ισραήλ να συμμετέχει στο Σικάγο. Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες δίκες στην Τουρκία, δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ να ασχοληθεί με εσωτερικά δικαστικά θέματα της Τουρκίας. Είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας και δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Κύριε Μπράντα, για την περιαγγελική άμυνα και το κόστος της έχω απαντήσει για την επικράτη που θα καλυφθεί από αυτό το σύστημα πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Θα καλύψει το ευρωπαϊκό έδαφος, το ευρωπαϊκό έδαφος χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι έχουμε προσδιορίσει την κάλυψη αυτού του νατοικού συστήματος πυραυλικής άμυνας. Έχουμε τη δυνατότητα να σας απευθύνουμε ακόμα τέσσερις σύντομες ερωτήσεις, ο καθένας σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Τους ακούμε όλους πρώτα. Ο Ποπόσκι είναι ο, το νούμερο 2 γενικός γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, και αν δεν μπορεί να μιλήσει, ε, θα ήθελα να έχουμε ακόμα δύο συνεδριάσεις ε, πριν το Σικάγο για να μπορέσει να μιλήσει. Για να δούμε και την άποψη της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Ε, ίδια ερώτηση με του Άντρου Νταφ. Αναφέρατε ότι οι ισχυρισμοί για το πραξικόπημα και τις ε, τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Τουρκία είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκία, αλλά σε αυτό επηρεάζει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ. Ε, και η διαδικασία και οι αποφάσεις των, οι τιμιγορίες των δικών αυτών ε, θα είναι σημαντικές για την αξιοπιστία της Τουρκίας. Ε, μήπως το ΝΑΤΟ θα στείλει παρατηρητές ούτως ώστε αυτές οι δίκες να γίνουν με βάση τα διεθνή πρότυπα και οι ισχυρισμοί που είναι πάρα πολύ σοβαροί δεν θα πλήξουν ανθρώπους αδίκως ε, ή αν αποδειχθούν αληθείς ε, να υπάρξουν οι απαραίτητες τιμωρίες, συνέπειες, κυρώσεις. Κύριε Πασκιού. Με την αναδιάρθρωση που υπάρχει στις ΗΠΑ Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι συνήθως ε, στην επερχόμενη Σύνοδο κορυφή. Πιστεύετε ότι οι σύμμαχοι συνειδητοποιούν την ανάγκη να υπάρχει κάποια αλλαγή πέρα από τα... την πεπατημένη. Υπάρχει περιθώριο να υπάρξει ένα νέο όραμα. Έχει το στρατηγικό δόγμα έχει υιοθετηθεί για τα επόμενα δέκα χρόνια βέβαια, αλλά υπάρχει περιθώριο για αυτό το νέο όραμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για την εσωτερική συνοχή της συμμαχίας, ειδικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την περιπολία στον ενέργειο χώρο της Βαλτικής. Επίσης για την επιχείρηση για τη Λιβύη. Για μένα η επιχείρηση στη Λιβύη είναι μαρτυρία του ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις στο εσωτερικό της συμμαχίας, της Νατοικής Συμμαχίας. Φυσικά καταλαβαίνω την άποψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, καταλαβαίνω την αισιοδοξία του, γι' αυτό σας πληρώνουν εξάλλου κύριε Γενική Γραμματέα. Αλλά δεν νομίζω ότι στρατιωτικά η επιχείρηση αυτά είναι και τόσο μεγάλη επιτυχία πια. Κύριε Γεωργίου. Καλώς ορίσατε κύριε Ρασμούσεν. Έχω τρεις μικρές ερωτήσεις. Άκουσα την ε, λαμπρή πραγματικά ανάλυση που έχετε κάνει για τα έξοδα ε, στα οποία μπαίνει η Ρωσία για την ανάπτυξη πυράβλων και τη θέση σας ότι θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να πάνε για κοινωνικούς ή ειρηνικούς σκοπούς και θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι πραγματικά αδύνατον να σκεφτείτε κάτι ανάλογο για τα έξοδα που κάνει το ΝΑΤΟ. Το δεύτερο που έχω να ρωτήσω, μετά τις εισβολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πιστεύετε ότι η ζωή των ανθρώπων εκεί έχει γίνει καλύτερη μετά από τόσες δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Το τρίτο αφορά την Ελλάδα, η οποία ξοδεύει ε, πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος για την άμυνα της. Ε, μπορεί το ΝΑΤΟ να κάνει κάτι για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την Τουρκία για να μειωθούν αυτοί οι εξοπλισμοί. Ε, έχω άλλε δύο μικρές ερωτήσεις. Εάν η Κύπρος κάνει αίτηση για ένταξη στο συνεταιρισμό, εσείς λέτε ή εγγυάστε για την στάση της Τουρκίας απέναντι σε αυτή την αίτηση. Και η τελευταία ερώτηση, ξέρετε καθόλου αν η Αγγλία έχει πυρηνικά όπλα στις βάσεις που έχει στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Για απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα. Ευχαριστώ προς την κυρία Σάκια καταρχήν. Όχι, είναι η απάντηση. Δεν είναι ευθύνη του ΝΑΤΟ να στείλει παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τις νομικές διαδικασίες, τις δίκες που λαμβάνουν χώρα στα μέλη του ΝΑΤΟ. Αν χρειαστεί, έχουμε άλλους διεθνείς οργανισμούς που μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση, λοιπόν, να στείλουμε νατοικούς παρατηρητές στην Τουρκία. Κύριος Πάσκου, με ρώτησε για τη σύνοδο κορυφής του Σάμιτ και το όραμα που μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να δείτε τη σύνοδο αυτή ως ε, το επόμενο βήμα και μια σύνοδο που θα συνεισφέρει στην εφαρμογή της, του στρατηγικού δόγματος που υιοθετήσαμε στη Λισαβόνα πριν από κάνα δύο χρόνια. Στο στρατηγικό αυτό δόγμα προσδιορίσαμε τα βασικά καθήκοντα του ΝΑΤΟ και στο Σικάγο θα τονίσουμε και θα προσδιορίσουμε τους τρόπους εφαρμογής αυτών. Και αυτό είναι τμήμα του οράματος. Το όραμα δεν είναι φλήνα φήματα. Το όραμα είναι κάτι απτό στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ακριβώς θα υιοθετήσουμε ένα αμυντικό πακέτο, όπως το λέμε, στο Σικάγο. Ένα πακέτο που πολύ απτά, πολύ συγκεκριμένα, θα δεσμεύσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για να επενδύσουν στο απαραίτητο στρατιωτικό δυναμικό τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας την έννοια της έξυπνης άμυνας. Θα είναι επίσης μια επανεπιβεβαίωση ε, στεναρή του διατλαντικού δεσμού. Και αυτό επίσης είναι τμήμα του οράματος του ΝΑΤΟ. Μπορεί η του Σικάγου να είναι πιο γιωμένη θα έλεγα έτσι, αλλά είναι τμήμα του οράματος. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο να έχεις όραμα και στο να μπορείς να εφαρμόσεις το όραμά σου. Το πιο εύκολο πράγμα εξάλλου είναι να είσαι θεροβάμωνας και να μιλάς για φοβερά όνειρα και οράματα και στόχους, αλλά δεν, δεν έχεις την ικανότητα, τον εξοπλισμό, τη δύναμη, τη θέληση να τα υλοποιήσεις, τι νόημα έχει. Η απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι το Σικάγο είναι τμήμα του οράματος και της εφαρμογής και υλοποίησης του οράματος. είπε ότι υπάρχει μια αντίφαση, μια διαφωνία ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και κυρίως εστιάσατε στην επιχείρηση της Λιβύης. Να σας διορθώσω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, όπως ξέρετε, όλες οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται ε, με συνένεση. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αναλάβει δεσμεύσει ε, απέναντι στη Λιβύη για αυτή την επιχείρηση χωρίς υποστήριξη και των 28 συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ίσως αυτό που υπενήσεστε είναι ότι δεν συμμετείχαν ενεργά ίσως όλες οι, όλες οι συμμαχικές χώρες στην επιχείρηση της Λιβύης. Ορισμένοι δεν έχουν τον εξοπλισμό, το δυναμικό για τέτοια επιχείρηση. Άλλοι δεν συμμετείχαν για άλλους λόγους. Αλλά και 28 σύμμαχοι υποστήριξαν την επιχείρηση και συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουμε το κοινό νατοϊκό πλαίσιο, την διοικητική δομή για αυτή την επιχείρηση. Η επιχείρηση της Λιβύης ήταν μια καθαρή απόδειξη ενότητας και αλληλεγγύης μέσα στη συμμαχία μας. Και στρατιωτικά ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ε, εφαρμόσαμε την εντολή του ΟΗΕ για προστασία του άμαχου πληθυσμού της Λιβύης. Αποφύγαμε την ασφαγή, αποτρέψαμε τη σφαγή και το πετύχαμε με έναν τρόπο όπου ε, ελαχιστοποίησαμε στο ελάχιστο δυνατό τις απώλειες των αμάχων και τις παράπλευρες απώλειες. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Κύριε Χατζηγεωργίου, ελπίζω, λέει ο μιλητής, να προφέρω σωστά το όνομά σας. Με ρωτάτε αν βελτιώθηκε η ζωή στο Αφγανιστάν. Ξέρουμε βέβαια ότι το Αφγανιστάν είναι μια κοινωνία με πολλές προκλήσεις, είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και μπορώ να σας πω ότι με αυτό το δεδομένο υπάρχει πρόοδος, πολύ πρόοδος. Πέρυσι νομίζω, η οικονομική ανάπτυξη ε, στο Αφγανιστάν ήταν περίπου 8%. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ε, υπάρχουν τρομερές βελτιώσεις 7 με 8 παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Εκατομμύρια παιδιά πηγαίνουν ε, στο σχολείο. Το 1 τρίτο είναι, τα, είναι κορίτσια από αυτά. Στο παρελθόν δεν είχαν το δικαίωμα να βάλουν το πόδι τους ε, στα σχολεία. Υπάρχει πρόοδο στην υγεία. Πολλά νέα κέντρα υγεία έχουμε στο Αφγανιστάν. Ε, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωή στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μείωση τη νησιμότητα των παιδιών. Έχουμε κατασκευάσει χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων νέων δρόμων που συνεισφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα, ε, ανοίγουν νέες αγορές στο Αφγανιστάν. Το, τα ΜΜΕ είναι έτσι πολύ δραστήρια στο Αφγανιστάν. Ναι, η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. Αλλά αν υπάρχει βελτίωση, η απάντησή μου είναι ε, έναν επιφύλακτο ναι. Υπάρχει βελτίωση. Τέλος. Για την Τουρκία και την Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν, υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αλλά το καλό είναι ότι χάρη στην Νατοική Συμμαχία, όπου συμμετέχουν και οι δύο χώρες, Αυτή τη στιγμή ε, εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, καταφέραμε να αποτρέψουμε, να λύσουμε αυτές τις ε, κρίσεις με ειρηνικό τρόπο. Και αυτό είναι που μετράει. Άλλο ένα, συν, ε, στις, άλλο ένα κρατούμενο στις επιτυχίες της ε, Ότι τέτοιες εσωτερικές διαφωνίες, διαμάχες επιλύονται με ειρηνικό τρόπο. Και οι δύο χώρες είναι ισχυροί σύμμαχοι και συνεισφέρουν με πολύτιμο τρόπο στις ανατολικές επιχειρήσεις. Και είναι προφανές ότι η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του πολιτισμού της και της θρησκείας της, παίζει ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό ρόλο. Ευχαριστώ κύριε Άντερς. Ε, θυμόμαστε την εποχή της Πρωθυπουργία σας. Ε, ήσασταν πολύ επιτυχής Πρωθυπουργός και τώρα αυτή την εμπειρία ε, τη δίνετε στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ηγεσία, νομίζω ότι μας βοηθάει όλους. Μα θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και κάποια σημεία που θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σχέση δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ίσως θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Και εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου μπορούμε να υποστηρίξουμε επικοδομητικά και να υποστηρίξουμε τα, τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να βελτιωθεί η σχέση ε, με τον ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι και σημαντικό για να εξοικονομήσουμε και χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Να έχουμε μια τέτοια κοινή προσέγγιση, γιατί μια τέτοια συνέργεια θα μας κάνει και ισχυρότερους, ε, θα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια, και ειρήνη και ελευθερία. Και θα το κάνουμε αυτό μάλλον, μάλιστα με τρόπο αποδεκτό ε, από όλους τους πολίτες. Καλή επιτυχία για το Σικάγο και ελπίζω να είναι πολύ πετυχημένη αυτή η σύνοδος. Πάμε πίσω στο σημείο 3. Θα καταγραφεί αυτό βέβαια και στα πρακτικά, αλλά το Σαββατοκύριακο έγινε μία διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρέθηκε ομοφωνία, συνένεση για την δημιουργία μιας διάσκεψης ε, της, ε, ε, για, για την ε, παρακολούθηση, αξιολόγηση της κοινή πολιτικής άμυνας. Δεν περίμενα ότι θα τα καταφέρναμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός συμβιβασμός μεταξύ όλων των συμφερόντων που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό θα γίνει δυνάμει του άρθρου 9 του πρωτοκόλου 1 για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε σημαίνει ότι η, ε, αυτό το, αυτή η συμφωνία θα είναι αντικείμενο των ε, Επιτροπών ε, Άμυνα και Ιστορικών Υποθέσεων, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν έξι εκπρόσωποι από κάθε κοινοβούλιο, 16 από το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Θα υπάρξουν και κάποιοι παρατηρητέ από τι υποψήφιε χώρε και από τα κράτη του ΝΑΤΟ που είναι μέλη της Ευρώπης, αλλά και για τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ευρώπης. Υπάρχει μια γραμματεία που αποτελείται από την Προεδρία από, το, από την Προεδρία που έχει τώρα δηλαδή την Προεδρία της Ένωσης και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προεδρεύει αυτής της ε, Επιτροπής. Θα είναι λοιπόν η καθήλια αρμόδια, ε, η Προεδρία αυτή θα είναι σε στενή συνεργασία βέβαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να παρακολουθούμε ε, στενά ε, το τι θα διαμειχθεί σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις. Θα υπάρξουν συνεδριάσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στη χώρα της Προεδρίας Δεν θα κάνουμε όλε τι συνεδριάσει βεβαίω στη χώρα τη Προεδρία γιατί είναι αρκετά δαπανηρό. Θα κάνουμε κάποιες από τι συνεδριάσει και εδώ στο Κοινοβούλιο και βεβαίω θα σα ενημερώνουμε ε, για το τι θα συμβαίνει. Ούτω ή άλλω υπάρχουν ε, ε, και συνάδελφοι οι οποίοι είναι μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και είναι μέλη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άμυνα και ασφάλεια Το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είχαμε πει ότι θα υπάρξει μετά από δύο χρόνια μία αξιολόγηση και θα δούμε, θα κάνουμε κάποιες συνεδριάσεις, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Στο τέλος βεβαίως θα υπάρξουν κάποια συμπεράσματα, δεν θα είναι δεσμευτικά, θα είναι συμπεράσματα επί της αρχής. Δηλαδή θα υπάρξει μια ενημερωτική ας πούμε ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την γραφειοκρατία που υπάρχει στα, στις χώρες μας. Πραγματικά αυτή η δυνατότητα μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια στενή σχέση μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να... Δεν θα αλλάξουν βεβαίως οι αρμοδιότητες, είναι σαφείς οι αρμοδιότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά αυτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν θέλουμε να ε, αναμειχθούμε ο ένας στα χωράφια του άλλου θα παραμείνουν οι ευθύνε όπως έχουν. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι που καταφέραμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την έργαση αυτή. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Ακόμη μία ανταλλαγή απόψεων με τον ειδικό πρόσωπο και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, τον κύριο Σουζάτσκας. Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Πραγματικά έχετε περάσει πολύ έντονες στιγμές, πήγατε στην Καμπούλ, νομίζω γυρίσατε στις 15 του Απρίλη, οπότε μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Ακούσαμε βεβαίω και την άποψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή να μα πείτε και εσεί το τι γίνεται στο Αφγανιστάν, γιατί και με αυτόν συζητήσαμε εντατικά το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι τιμή μου που μπορώ να απευθυνθώ σήμερα ενώπιόν σα, ε, Μετά από την παρουσίαση βεβαίως και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τι δικέ μου απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο Αφγανιστάν. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελευταία δεκαετία η διεθνής κοινότητα και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχουν κάνει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των κοινών στόχων της, της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της δημοσιονομικής εξυγένσης στο Αφγανιστάν και την παροχή ασφάλειας στους, στους Αφγανούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία είναι πραγματικά πρωτοφανή, Η ποιότητα και η ποσότητα των ε, δυνάμων ασφαλείας συνεχίζει να αυξάνεται στο Αφγανιστάν. Η ασφάλεια στον, σε πολλές πόλεις έχει βελτιωθεί, ειδικά στο νότιο Αφγανιστάν. Περίπου μισή από τον, το 50% του πληθυσμού είναι στην ε, αρμοδιότητα των δυνάμεων ασφαλείας. Πραγματικά το Αφγανιστάν είναι μια πολύ δύσκολη χώρα. Η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. Είδαμε τι έγινε και με τις επιθέσεις στην Καμπούλ την προηγούμενη εβδομάδα οι γυναίκες πραγματικά δεν βρίσκονται καθόλου κοντά στο να έχουν μια ίση θέση στην κοινωνία. Η ε, βιωσιμότητα λοιπόν όλων αυτών των ε, στόχων που έχουμε πετύχει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια έχει να κάνει και με το πώς θα το παρακολουθήσουμε και θα έχουμε καλή διαχείριση. Αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική διαχείριση αλλά και, τα, για τα θεσμικά όργανα της χώρας για να υπάρξει πρόσβαση στην δικαιοσύνη και να υπάρξει επίτευξη των στόχων για την, ε, για την προσέλκυση επενδύσεων και να υπάρχει, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Ε, η, συνεργασία λοιπόν είναι σημαντική για να μπορέσει αυτό να διατηρηθεί στο Αφγανιστάν και στη γενικότερη στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική για την υποστήριξη της Αφγανικής κυβέρνησης ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και να υπάρξει ευημερία. Με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δέσμευση των αφγανικών αρχών, αυτή η στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει. Οι επόμενες διασκέψεις στο Τόκιο, το Σικάγο και την Καμπούλ φέτος δίνουν μια δυνατότητα έτσι ώστε αυτές οι ανθρώπινες και οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο Αφγανιστάν να δημιουργήσουν ε, θεμέλια έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στο μέλλον. Θα θυμάστε ότι στη Βόνη τον προηγούμενο Δεκέμβριο η διεθνή κοινότητα ε, επιβεβαίωσε την δέσμευσή της για την ενίσχυση του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης που θα υπάρξει στη χώρα μετά το 2014. Επίσης, η αφγανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να κάνει την ε, διάσκεψη στο, στην Καμπούλ για να ενισχυθεί το κράτος δικαίου, οι ε, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ε, ώστε να, υπάρξει, να υπάρξουν καλύτερες ε, προοπτικές για ε, διεθνείς επενδύσεις, για ανάπτυξη και για οικονομική ευημερία. Από την ώρα που ελήφθη η απόφαση πέρσι από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και από την ύπατη εκπρόσωπο Κάθι Άστον, υπάρχει σαφής δέσμευση να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση για το Αφγανιστάν και για την ευρύτερη περιοχή και διμερώς αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευρυνθεί αυτή η ανάπτυξη και να ε, διευρυνθεί και η εντολή της Γιούπολ έτσι προσέχοντας βεβαίως να υπάρχει σαφής, ε, ε, σαφές κράτος δικαίου, ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων μετά το 2014. Η διεθνή κοινότητα πραγματικά αποδίδει μεγάλη σημασία στην, στις διασκέψεις αυτές. Η διάσκεψη του Τόκιο θα επικεντρωθεί στην διακυβέρνηση Προσπαθούμε να ε, τονίσουμε και την δέσμευση του Αφγανιστάν και την ε, ε, στρατηγική που έχει εκπονηθεί, έτσι ώστε το Αφγανιστάν να μπορέσει να είναι αυτόνομο. Είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές η, περιοχή, η ευρύτερη περιοχή του Αφγανιστάν, οπότε θέλουμε προφανώς να ενισχύσουμε την ευημερία των πολιτών. Το Αφγανιστάν συνδέει την Κεντρική, την Νότια Ασία, την Ευρασία και την Μέση Ανατολή. Έχει, είναι πλούσιο σε χαλκό, χρυσό και σίδηρο. Έχει λοιπόν πολλούς, πολλές πρωτοπαραγωγικές πηγές, αλλά το Αφγανιστάν για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όλα αυτά χρειάζεται ε, υποστήριξη. Και αυτό βεβαίως ε, επιβεβαιώθηκε και από μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο Τόκιο περιμένουμε ότι η Αφγανική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την δέσμευσή της να ε, υποστηρίξει τις δεσμεύσεις στην Καμπούλ σε ό,τι αφορά κυρίω τη διακυβέρνηση και σε ό,τι αφορά την ε, κυβέρνηση, όντω πρέπει να, γίνει, ε, να αναλυφθούν δράσει έτσι ώστε το Αφγανιστάν να διατηρήσει την ε, υποστήριξη και του δικού σα κοινοβουλίου αλλά και των πολιτών και των κρατών τη Ευρώπη. Και αυτό θα, σημαίνει μια αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα, ώστε να υπάρξουν επιπλέον επενδύσεις και στην οικονομική και στην κοινωνική ανάπτυξη με πιο συντονισμένο τρόπο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα εθνικά προγράμματα τα οποία έχουν προκύψει μετά από την διαδικασία της Καμπούλ και ταυτόχρονα η διεθνής κοινότητα ε, θα επαναλάβει την ανάγκη για σωστή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την στρατηγική αυτή που θα αντικατοπτρίζει και τη δυνατότητα απορρόφησης τη ε, αφγανική κυβέρνηση, αλλά και τα μειούμενα επίπεδα βοήθεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την βιωσιμότητα των εθνικών δυνάμεων ασφάλεια στο Αφγανιστάν. Οι αρχές έχουν συμφωνήσει να ενισχύσουν τις ε, δυνάμεις αυτές και να φτάσουν το 228.000 σε προσωπικό με μια πρικοδότηση 500 εκατομμύρια για, παρόλο που το κόστος αυτής της ε, όλης ε, επιχείρησης είναι ένα δις το χρόνο. Η ευρωπαϊκή λοιπόν χρηματοδότηση για την, ε, ε, ευρωπαϊκή, για την αφγανική συγγνώμη, αστυνομική, αστυνομικές δυνάμεις ε, θα διαρευνηθεί από το 2014 και τα λοιπά όταν θα λήξει και η εντολή. Η σταθερότητα και η ανάπτυξη στο Αφγανιστάν εξαρτώνται από την υποστήριξη των, περιφερειακών, των, των γειτονικών κρατών. Πρέπει λοιπόν να προωθηθεί ε, και η περιφερειακή ανάπτυξη και μετά την ε, διάσκεψη στην ε, Κωνσταντινούπολη και η αυγανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τη για συνέχιση τη συνεργασία και την ανάληψη τη ευρωπαϊκή βοήθεια για καλύτερη συνεργασία. Προς το παρόν οι χώρες της καρδιάς της Ασίας όπως λέγονται ε, προσπαθούν να, προβλέπ, να προετοιμάσουν τέτοια μέτρα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, για τη συνεργασία, για την διαδραστικότητα και για την αντιμετώπιση των, ε, του, του λαθρεμπορίου. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα και με το πρόγραμμα δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση των ε, αφγανικών δυνατοτήτων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, την, ε, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, τη ε, περιφερειακή συνεργασία και των δυνάμεων ασφαλεία. Έχει υπάρξει πρόόδο. Ε, συμπεριλαμβανομένη ε, και τη βοήθεια βεβαίως που έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταρρύθμιση των ε, διοικητικών δομών. Α πούμε, η δημόσια υγεία. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και αυτό έχει συμβάλει στο να υπάρξει ένα Υπουργείο υγεία. Επίση, τα προγράμματα περιφερειακή ανάπτυξη προωθούνται από τα σχετικά Υπουργεία. Βεβαίω υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δυνατο... δημιουργία δυνατοτήτων. Προφανώ υπάρχουν ακόμη μεγάλε προκλήσει. η πρόοδος ε, για, ε, για τη διακυβέρνηση της χώρας εξακολουθεί να είναι ε, μικρή. Η μεταρρύθμιση ό,τι αφορά την, τις εκλογικές διαδικασίες στη χώρα είναι σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο πρόεδρος Καρζά έχει αναφέρει ότι θέλει να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση και να γίνει άμεσα. Φέτος, ο, τώρα αυτό το μήνα, συγγνώμη, έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος να υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου και μάλιστα προχτές έγινε η πρώτη δημόσια διαβούλευση για τις προτινόμενες τροπολογίες για τον εκλογικό νόμο. Όλα αυτά έγιναν στην Καμπούλ. Αυτό ο διάλογο λοιπόν είναι σημαντικό ε, γιατί στις, ε, το 2014 θέλουμε να είναι διαφανεί και ελεύθερε οι εκλογέ που θα γίνουν και αυτό να το καταλάβουν και οι Αφγανοί. Επίση, το ο Αφγανιστάν προσπαθεί να δημιουργήσει μια κοινοβουλευτική παράδοση. Η ευρωπαϊκή κοινότητα πρέπει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Οπότε θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί ε, μεταξύ των ε, σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Εθνικό Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προγραμμάτων για την, για την ε, ενίσχυση των δυνατοτήτων αλλά και τη δημιουργία μιας πολιτικής κουλτούρας. Η βιώσιμη ειρήνη στο Αφγανιστάν είναι συνεχιζόμενη μέσω ενός συστήματος πάνω στο οποίο θα μπορούν όλοι οι ε, Αφγανοί να έχουν τα ίσα δικαιώματα. Και βεβαίως θέλουμε και τη συνεργασία με, τον, ε, με τη γειτονική χώρα, το Πακιστάν. Τον Ιανουάριο φέτος ε, υπήρξε νέα δυναμική γιατί για πρώτη φορά η πακιστανική κυβέρνηση ήρθε, έκανε έκκληση στους Ταλιμπάν να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Υπάρχει λοιπόν ετοιμότητα από τους Αφγανούς και από τους Πακιστανούς να δημιουργηθεί μια διαδικασία ειρηνευτική και αυτό βεβαίω είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Παρ' όλα αυτά, όπω ξέρουμε όλοι, η σχέση μεταξύ των Ταλιμπάν και των ε, Πακιστανών είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι Ταλιμπάν όντω θα, ε, θα έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Καμπούλ. Ο κύριος Ραμπάνη πριν από δύο ε, μέρες ανέφερε ε, ότι ε, επιβεβαίωσε μάλλον την ε, δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τόνισε την ανάγκη που υπάρχει να εξασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι συνεπέ με, με τα διεθνή πρότυπα και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει πολιτικά το πρόγραμμα ολοκλήρωσης και ειρήνης στο Αφγανιστάν, στο και πρέπει να ενισχύσουμε την, ε, τις δυνατότητες ε, ενσωμάτωσης που υπάρχουν, αλλά είναι λίγο ανησυχητικέ οι δυνατότητες που έχουν τα Υπουργεία να δώσουν τις ε, ευκαιρίες που υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρξει βιώσιμη διαδικασία ολοκλήρωσης. Για το κράτος δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει σημαντικά για να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση ώστε να προωθηθούν τα πολιτικά δικαιώματα και γιατί η στρατιωτική, η στρατιωτική ε, προστασία προφανώς είναι τελείως διαφορετική από την παραστρατιωτική, η οποία εξακολουθεί να έχει ε, ισχυρούς δεσμούς στη χώρα. Βεβαίω πρέπει και η διεθνή κοινότητα να ε, ενισχύσει την, ε, τις αστυνομικές δυνάμεις και την μεταρρύθμιση του αστυνομικού σώματος αλλά και του δικαστικού αυτό βεβαίω πρέπει να γίνει από κοινού με το Υπουργείο Ιστορικών στο Αφγανιστάν. Προφανώ ε, ε, υπάρχει ανάγκη για τεράστιε προσπάθειε για του δύο αυτού ε, τομεί και πρέπει να ενισχυθούν. Δυστυχώ η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει βελτιωθεί του τελευταίου μήνε στο Αφγανιστάν. Η διακριτική μεταχείριση και η βία κατά των γυναικών συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ ενισχυτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει την ε, στήριξή τη για την ε, κοινωνία των πολιτών και εξεκολουθεί να μιλά για την ε, αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν και των ελλείψεων σε ό,τι αφορά τα όσα κάνει η αφγανική κυβέρνηση. Για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με την Αφγανική ε, κυβέρνηση για να ενθαρρύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, για να υπάρξει ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα και στον ε, τομέα των εξορίξεων και να δημιουργηθεί ένα ε, εμπορικό επιμελητήριο στο Αφγανιστάν. Όλα αυτά θα, θα ωφελήσουν προφανώς την περιοχή, θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη στο Αφγανιστάν η πρόσφατη διάσκεψη που έγινε δείχνει ότι σε αυτό το περιφερειακό μέτωπο θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Στο Αφγανιστάν η ανθρωπιστική βοήθεια, έχει, οι ανθρωπιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί. Ε, είναι πολύ περιορισμένη πολλές φορές και ε, ανύπαρκτη η πρόσβαση κάποιων ε, τμήματων του πληθυσμού σε άλλα, σε άλλα σημεία της χώρας Προφανώ πρέπει να υπάρξει ε, προστασία των πολιτών, ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, έχουν ε, δοθεί περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για του ανθρώπου που πραγματικά πλήττονται από τι διαμάχε και από τι φυσικέ καταστροφέ. Και για του ανθρώπου που χάνουν τα σπίτια του. Προφανώ η ευρωπαϊκή βοήθεια στο Αφγανιστάν έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να αυξηθεί και η ασφάλεια και η ανάπτυξη στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω έχει ε, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή τη μεταρρύθμιση του Αφγανιστάν και κυρίω από, από το 2014 και μετά. Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία αυτή για την εταιρική σχέση και για την ανάπτυξη που ξεκίνησε το Μάρτιο φέτο και προγραμματίζεται και ένα δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μήνα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό και θα, γίνει, θα υπάρξει ένα ε, δεσμευτικό πλαίσιο για τι σχέσει με το Αφγανιστάν για τα επόμενα χρόνια που θα καθορίζει μια κοινή κοινή ατζέντα για κοινέ αξίες και υποχρεώσεις για τομείς όπως ε, ε, οι επενδύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και άλλοι. Κλείνοντας να πω ότι είναι σαφές ότι το Αφγανιστάν χρειάζεται περισσότερα, κάτι περισσότερο από την απλή ε, ασφάλεια για να αφήσει πίσω το 30 χρόνια πολέμου. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, βιώσιμο, μια βιώσιμη προσέγγιση που να ενισχύει τα, τις ε, διοικητικές δομές, να αντιμετωπίζουν τα, τα κενά που υπάρχουν, να ενισχύει τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε το οικονομικό πλαίσιο να ενισχυθεί για να υπάρξει την οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η, η διεθνή κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα μέσω ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ μα και με την αφγανική κυβέρνηση. Οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το πώ θα γίνει τελικά αυτό στην πράξη. Από το 2014 και μετά πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση από, ένα, από μια προσέγγιση ε, στρατιωτική σε μια προσέγγιση πολιτική. Θα φύγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις από τη χώρα το 2014 και το 2014 θα εξακολουθήσει να είναι το Αφγανιστάν μια χώρα από τις πιο φτωχές του κόσμου. Θα συνεχίσει λοιπόν να χρειάζεται διεθνή βοήθεια για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά όπως και άλλα παραδείγματα τέτοιων χωρών μας έχουν δείξει, τα κράτη πρέπει να βρουν το δικό τους δρόμο για να προχωρήσουν και να βρουν τους δικούς τους πόρους για να ενισχύσουν την ε, ανάπτυξή τους και να εγγυηθούν το ένα βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες τους. Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ, η διεθνής κοινότητα δεν μπορούν να κάνουν τα λάθη α, του, της δεκαετίας του 90 και να ε, γυρίσουν την πλάτη τους στο Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αν έχετε ερωτήσεις ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος από τη Ιταλική Βουλή. Κύριε εκπρόσωπε, Ποιο είναι ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2014. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη θέλει να αυξήσει την ε, ενεργοποίησή της, τη δραστηριοποίησή της υπέρ της ε, καλής διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών στο Αφγανιστάν. Δεύτερον, τι άποψη έχετε για τις πιθανές εξελίξεις της κατάστασης στο Ιράν. Και αυτό σε συνδυασμό με το Αφγανιστάν. Τρίτον, Ποια είναι η γνώμη σας για τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει μεταξύ της συμμαχίας και της κυβέρνησης ε, Καρτζάη και των Ταλιμπάν. Μπορεί να παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο ερώτημα. Από ευρω... πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια αξιολόγηση για το γεγονός ότι μετά το 2014 πρέπει να παρασχεθεί προστασία στους εκπαιδευτές. Και αυτή η προστασία των εκπαιδευτών πώς θα εξασφαλιστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι καλώς ορίζω θερμά τον κύριο ε, Ουζάσκατς εδώ στην Επιτροπή μας. Και βέβαια όλοι οι δύο ρωτούνται τι θα συμβεί με την ασφάλεια της χώρας και θα γίνουν τα έργα και τα μέτρα μας μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων το 2014. Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό τομέα, πιστεύω ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ και γενικότερα η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναμένει ότι μετά την αποχώρησή μας δεν είναι σε θέση κυβέρνηση, αν μη τι άλλο να φροντίζει, να μην ε, εξαπολύονται τρομοκρατικές απειλές από την αφγανική επικράτεια. Πράγμα που συνέβαινε στο παρελθόν. Τουλάχιστον ε, αυτό θα περίμενε κανείς ε, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Τώρα τα δικά μας έργα και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτώ. Πώς συνεργαζόμαστε με τους διάφορους πολιτικούς φορείς, την κυβέρνηση, τα κόμματα, τις φυλές. Συζητούμε τα μέτρα μας ε, με στόχο να δημιουργηθεί μια συνένεση. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε για την υγεία, για την παιδεία, για τις υποδομές, μπορούμε να επιτύχουμε όχι η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και κάποια επόμενη, είτε είναι αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού, είναι μια τελείως διαφορετική στη σύνθεσή της, θα το συνεχίσει αυτό. Ε, πώς κάνουμε εκεί το διάλογο, πέρα από τα νυν Υπουργεία με τους διαφόρους ενεχομένους για να εξασφαλίσουμε και μια διάρκεια και μια συνέχεια και μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων αλλά και από μια διαφορετική κυβέρνηση θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Αυτά που όντως κάνουμε και επενδύουμε για τον κόσμο οι στοδυνικές θα συντηρηθούν, θα αναγνωριστούν από τους ηθήνοντες. Ευχαριστώ. się złożyło, że w ciągu ostatnich lat e, bardziej patrzyłem ε, na Μετά από τόσα χρόνια παρουσία στο Αφγανιστάν θα πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό και από τη σκοπιά του ΝΑΤΟ και από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω υπολείπεται κατά πολύ των δυνατοτήτων που θα είχε. Ας πούμε, η Συμμαχία έχει επιλέξει μια συνολική προσέγγιση Δηλαδή και στο Αφγανιστάν αλλά και σε άλλες ε, περιοχές υπάρχει πρόθεση στρατιωτικής παρουσίας. Αλλά όχι μόνο. Είναι και αναπτυξιακή βοήθεια και η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν καλό και σκόπιμο να το επομιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά το 2014 θα είναι ακριβώς ε, κρίσιμη η καμπή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ρόλο και ενδεχομένως να χρειαστεί να παραμείνουμε στην Κεντρική Ασία. Και να ρωτήσω κάτι. Αυτό τον καιρό επίκειται ένας τρίτος γύρος παράδοσης ε, σε διάφορες περιοχές ε, και επαρχίες. Στους δύο προηγούμενους γύρους είδαμε ότι η παράδοση γινόταν με επίσημο τρόπο, με τελετές, αλλά και μετά από κάποια πολιτική επιρροή. Ε, Μπαμιάν Παντσίρ Μασάρελ Σαρίφ ήταν στον πρώτο γύρο η παράδοση και αυτά έγιναν με βάση κάποια κριτήρια. Ενώ οι δύο άλλες πόλεις που ακολούθησαν ήταν αμυγός πολιτική πράξη. Και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Ουσάτσκας, στο μέλλον τι θα γίνει. Γιατί όσο περισσότερο παίρνονται πολιτικές αποφάσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αστάθεια ε, στο μέλλον. Μειώνεται η σταθερότητα της χώρας. Και ένα τρίτο, εν ώψη και των συζητήσεων που κάναμε μάλλον προηγουμένως με το Γενικό Γραμματέα του ε, ΝΑΤΟ. Έχω μια ερώτηση για το δεύτερο ήμιση του 2013 και το 2014. Τι σημαίνει όταν λέγει η διεθνής κοινότητα ότι το ΝΑΤΟ θα περιορίσει τη δράση του σε υποστηρικτική δράση. Τι σημαίνει αυτό. Η συμμαχία θα υποστηρίζει τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Με ποιο τρόπο. θα περιοριστεί η στρατιωτική μας παρουσία εκεί και η δράση μας, αλλά αυτό μπορεί ενδεχομένω να σημαίνει μεγαλύτερη απειλή. Αν αυτή η απόφαση ληφθεί στο Σικάγο, γιατί από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο θα γίνει, ποιες θα είναι οι στρατιωτικές συνέπειες, τις έχουμε σκεφτεί, ποια ε, είναι, ποιο σκοπό, στρατιωτικό σκοπό εξυπηρετεί μια τέτοια δήλωση. Τι σημαίνει υποστηρικτική δράση του ΝΑΤΟ εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Υποστηρίζουμε τι αφγανικέ δυνάμει Με ποιο τρόπο. Η κυρία Κοπά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω τρει πολύ σύντομε ερωτήσει. Πρώτον, για το ρόλο τη Εθνική Αστυνομία στο Αφγανιστάν. Ο ρόλο τη, μετά την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων ποιο θα είναι. Γιατί ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και κάποια από τα πιο βασικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι αστυνομικοί δεν υπάρχουν. Βασικά προβλήματα είναι η διαφθορά, ε, η αγραμματοσύνη και η διατροφή του πληθυσμού. Μετά την αποχώρησή μας το 2014 είναι πιθανόν οι, τα αντάρτικα να αναζωπηρωθούν. Τι ρόλο θα έχουν λοιπόν οι αστυνομικέ δυνάμεις σε αυτή τη φάση. Δεύτερο, ε, κάποιες παλιές επικρίσεις για το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λόγω των, διαφορετικών αρμοδιότητων που έχουν, έχουν οι διάφοροι φορείς. Ε, και επιπλέον διάφορα κρατημέλη έχουν διαφορετικές απόψεις για το Αφγανιστάν ο εσωτερικός ε, ευρωπαϊκός συντονισμός πώς ε, θα αλλάξει τώρα που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και πώς θα αναπτυχθεί στο μέλλον ο συντονισμός αυτός. Τελευταίο, για τις πρόσφατες επιθέσεις που έγιναν από Ταλιμπάν και Αντάρτες ε, ταυτόχρονα σε διάφορα, διάφορες περιοχές στο Αφγανιστάν και στην πρωτεύουσα την Καμπούλ και στη λεγόμενη πράσινη ζώνη. Προφανώς αυτό ήταν απόδειξη ισχύω των ομάδων αυτών. Υπάρχει και μια απόπειρα να αμφισβητηθεί η ετοιμότητα των αφγανικών δυνάμεων για να αναλάβουν ε, την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας στο μέλλον. Με δεδομένο αυτό, είναι οριστικό ότι μια απλή στρατιωτική λύση στο πρόβλημα των Ταλιμπάν δεν είναι δυνατή και πρέπει να διερευνήσουμε και διπλωματικές οδούς. Έχουμε κάποια στρατηγική γι' αυτό. Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική. Θα πρέπει να συνδυάσουμε στρατιωτικά μέσα και διπλωματικές προσπάθειες και ποια είναι τα βήματα που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ και βουνομονώ ε, το Βιγιούντα τον πρέσβη Ουσάσκας. Διακινδυνεύετε ε, η ζωή σας κάθε μέρα και τη δική σας και της οικογένειάς σας στην Καμπούλ και στην περιοχή και σας ευχαριστώ που το κάνετε αυτό για τα ιδανικά και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σπουδαία η αποστολή σας και την εκτιμούμε βαθύτατα. Δεύτερο, μια που μιλούμε για τις αξίες που εκπροσωπείτε εσείς εκεί, οι αξίες μας οι οποίες βασίζονται στη γαλλική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ή την οικουμενική διακήρυξη των Ηνωμένων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα πρώτα θεμέλια για μια στοιχειώδη κοινωνία των πολιτών. Μετά όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε στην αφγανική κοινωνία, πώς αξιολογείτε την κατάσταση, ποια είναι η διαφορά από τότε που πρωτοπήγατε μέχρι σήμερα, πόσο μεγάλη ήταν η πρόοδος και πώς βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι η κοινωνία λιγότερο ε, φονταμεταλιστική, να μην βασίζεται τόσο πολύ στο μίσος και να προσανατολιστεί περισσότερο στα πολιτικά δικαιώματα, τα αστικά δικαιώματα, γυναικεία δικαιώματα και γενικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μπορείτε με δύο λόγια να μας περιγράψετε. Ε, όχι τη στρατιωτική πραγματικότητα, την πραγματικότητα των ε, αξιών μας, η κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράσμουσεν προηγουμένως μας μίλησε για το μέλλον ε, της δέσμευσης του ΝΑΤΟ για τις εκπαιδευτικές αποστολές και τα λοιπά στο Αφγανιστάν. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το μέλλον της Γιούπολ στο Αφγανιστάν. Ποιος είναι ο ρόλος εκεί ε, της αποστολής μας, θα συνεχιστεί καν και με ποιες προϋποθέσεις θα ενταχθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αποστολών που έχει τη διοίκηση το ΝΑΤΟ. Ποιο είναι ο ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ο κύριο Ράσμουσεν μα είπε ότι οι εκπαιδευτικέ αποστολέ θα πρέπει να έχουν και μια στρατιωτική εξασφάλιση και κάλυψη. Εκεί πώ βλέπετε εσεί το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε σκεφτεί επίσης και κάποιες τάξεις μεγέθους, να μας δώσετε και αριθμητικά στοιχεία σε περίπτωση που συνεχιστεί η αποστολή γιου εκπαιδευτική και αυτή της Ένωσης. Γιατί στην αρχή ακούσαμε ότι μέχρι, ε, μέχρι τα τέλη του 12 θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 352.000 ε, στρατιωτική και αστυνομική στο Αφγανιστάν. Μετά μειώθηκε αυτός ο αριθμός και έγινε 230.000. Σήμερα σε ποια επίπεδα κινείται. Έχω κι εγώ ερώτηση, ε, Πρόεδρος. Αναφέρθηκε και το αναφέρετε και εσείς η επιρροή του Πακιστάν και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και πολιτικά. Γιατί το Πακιστάν έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια την ίδια του Αφγανιστάν. Συνεργασία μεταξύ του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και των συμμαχικών δυνάμεων. Θα συναντηθούμε και με τον γεωργιστή Ραμπάνη, δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε τίποτα από αυτά για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ ε, όλα τα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το Αφγανιστάν και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και την υποστήριξη στο φίλο μου, τον Ζίγκερης. Ε, πραγματικά είμαι μόνος μου στην Καμπούλ. Η μετάθεσή μου εκεί δεν αφορά και την οικογένειά μου. Είμαι μόνος στην αποστολή αυτή και ε, εκτελώ τα καθήκοντά μου σε ό,τι αφορά ε, ε, όσα ρώτησε ο κ. και η κυρία Λόιζεκ, ποιος είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2014 και της Ιούπολ. Νομίζω, με κάθε συμβασμό, ε, άκουσα και τον Γενικό Γραμματέα Ράσμουσεν όταν σκιαγράφησε λίγο τις σχέσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά με όλο το σεβασμό πιστεύω ότι δεν θα ήταν ε, σωστό να το περιορίσουμε μόνο στην εργασία της ISAF με τη UPOL. Είναι πολύ ευρύτερη η δέσμευση εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρουσία στο Αφγανιστάν μαζί με τον ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς ε, φορείς. Και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις αλλά 30.000 Ευρωπαίοι πολίτες μοιράζονται αυτό το βάρος με τους Αμερικανούς και με άλλους στο Αφγανιστάν. Είμαστε μεγάλους ζωητής ανθρωπιστικής βοήθειας. Γνωρίζετε, η USAID έχει ένα προϋπολογισμό για φέτος 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια η Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη και τον κοινοτικό προεπολογισμό ε, δίνει ένα δισεκατομμύριο περίπου. Δηλαδή έχουμε, να πούμε πολλά, έχουμε μεγάλο λόγο και στο πολιτικό πεδίο, όχι μόνο στο αναπτυξιακό. Η αστυνομική μας αποστολή επίσης ε, αυξάνεται σε σημασία και πριν από δύο χρόνια όταν έφτασα στο Αφγανιστάν ήταν, είχαν αρνητική εικόνα για τη Γιούπολ. Όχι μόνο ε, ηθήνοντες εκεί του Αφγανιστάν αλλά και σε κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης. Τώρα η Γιούπολ αυξήθηκε σε σημασία και προβολή πάρα πολύ διότι έδειξε η κατάσταση επιτόπου ότι χρειάζεται εκπαίδευση η αστυνομία ε, αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς, εκπαιδεύουμε αστυνομικού και κανείς άλλος ε, από τους διεθνείς φορείς δεν μπορεί να παρέχει αυτή την εκπαίδευση. Απαντώ λοιπόν σε διάφορες ερωτήσεις που έγιναν για το μελλοντικό μας ρόλο, λέγοντας το εξής. Όπως σας είπα, 27 Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν τον Νοέμβριο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρική σχέσης και σύνδεσης που είναι νομικά δεσμευτική και είναι συνολική η συμφωνία. Καλύπτει πολλούς τομείς και τουλάχιστον αφορά την επόμενη δεκαετία. Ε, αυτή η συμφωνία θα χαράξει και ένα οδικό χάρτη για τη μελλοντική συνεργασία της Ένωσης και των 27 κρατών και των Αφγανιστάν. Ανθρώπινα δικαιώματα, εμπόριο, περιφερειακή συνεργασία, επενδύσεις, ε, δημιουργία δυνατοτήτων, ε, ικανοτήτων και αστυνομία δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα της Γιούπολ. Σήμερα το πρωί, ε, μόλις έφτασα, ε, με τους συναδέλφους στις διάφορες επιτροπές, CPC και CPMD. Γίνεται αυτό τον καιρό μια στρατηγική αναθεώρηση της Γιούπολ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι το πιθανότερο. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μονομένοι, απομονωμένοι παίκτε εκεί. Θα πρέπει να τα δούμε σε ένα συνολικότερο πλαίσιο και ποιο θα είναι το γενικότερο αποτύπωμα που θα αφήσει η διεθνή κοινότητα. Ακούσαμε τον κύριο Ράσμουσε να λέγει ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει και μετά το 2014 παρουσία και μια εκπαιδευτική αποστολή. Και όπω ρώτησε και ο Μίχαελ Γκάλερ, ποιο θα ε, ε, εξασφαλίζει εκεί την ασφάλεια των διαφόρων προγραμμάτων που έχουμε εμείς αυτόν τον καιρό και αυτό θα πρέπει να απαντηθεί σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και όλο και περισσότερο τους περιφερειακούς εκεί εταίρους. Ε, ακούστηκε η δυναμική Ιράν-Αφγανιστάν. Για να είμαι ειλικρινής, στην Καμπούλ έχω καλές σχέσεις εγώ με τους Ιρανούς και τον Ιρανό πρέσβη. Ενδιαφέρονται πολύ να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνούς παράγον, παράγοντες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών κυρίως. Συμμετείχα πριν από δέκα μέρες σε μια διάσκεψη προκαταρκτική στην Ασραμπάτ για την επερχόμενη περιφερειακή διάσκεψη στην Καμπούλ, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Καζαχστάν και Ινδία εξέφρασαν ενδιαφέρον να ε, προεδρεύσουν σε μια ομάδα εργασία. Για μα λοιπόν είναι φυσικά αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα και μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα επικοδομητικό ρόλο αντιμετωπίζοντας περιφερειακές προκλήσεις μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους. Διαπραγματεύσεις ρωτήσατε του Καρζάη με τους Ταλιμπάν. Ναι προδεκαημέρου αν δεν απατώμε στις 16, όχι, 15-16. Πότε ήταν ε, οι επιθέσεις στις 14, πριν τις επιθέσεις, στις 14 Απριλίου ε, ήρθε μια αντιπροσωπεία του Βισλάμι και ε, επισκέφθηκε την Καμπούλ και είχαν συζητήσεις με την κυβέρνηση. Ο κύριος Ραμπάνη που μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ε, τους ε, παρέθεσε ε, γεύμα εργασίας. Έχουν κάποια αιτήματα, τουλάχιστον μία ομάδα διαπραγματεύεται άμεσα με την κυβέρνηση Καρζάη. Μέρη νομίζω απάντησα για το τι θα γίνει με την ασφάλεια των εκπαιδευτών. Επίσης ρώτησε ο Μίχαλ Γκάλερ για τη διάδραση και συνεργασία με ένα ευρύτερο φάσμα ε, της αφγανικής κοινωνίας. Ε, ε, ουλεμάδες, διάφοροι περιφερειακοί ηγέτες, φύλαρχοι. Μίχελ, σε τακτά χρονικά διαστήματα βλέπω εκπροσώπους από το Κανταχάρ, από τον Νότο Ανατολή, Δύση, όχι μόνο εγώ και άλλοι εκπρόσωποι της Ένωσης και των κρατών μελών Καταλαβαίνετε ότι δεν συνεργαζόμαστε μόνο με την κυβέρνηση, δεν πρόκειται γι' αυτό. Είναι πολύ περίπλοκη η δομή της κοινωνίας στο Αφγανιστάν. Έχει τις δικές της παραδοσιακές δομές και τρόπους ε, λειτουργίας και business κάνουν με πολύ ε, απάνθρωπο τρόπο, έτσι, απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να αναπτυχθεί η κοινωνία. Και ε, Μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου, γιατί έχω δεχτεί διάφορες αντιπροσωπείες, είτε μέλη επαρχιακών συμβουλίων, είτε ε, πηγαίνοντα στην Παρασκευή στη Σούρα και πρώην ηγέτες των Ταλιπάν που έχω συναντήσει στην Καμπούλ, έχω αποκομίσει την αίσθηση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ε, χώρα πιάνει τόπο. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση του κυρίου Κλίχ για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν φαίνεται να συνεργάζονται, να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Νομίζω ότι είναι σφάλμα αυτή η εντύπωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις η συζήτηση επισκέζεται από τη στρατιωτική πτυχή. Εμείς είμαστε βαθύτατα δεσμευμένοι και προσιλωμένοι στην ανάπτυξη ιδρυμάτων και, και μάλλον όχι, στην ανάπτυξη θεμελίων ενός κράτους ε, που θα είναι πραγματικό κράτος και θα ζει ειρηνικά στην επικράτειά του και θα συνεπάρχει ειρηνικά με τους γείτονές τους. Θα αλλάξει σημαντικά η κατάσταση μετά το 2014 όταν φύγουν τα στρατεύματα. Για να απαντήσω και στην ώρα της κυρίας Κοπά, Θα παραμείνουμε και μετά το 2014. Είμαστε δεσμευμένοι όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Εξού και οι επικείμενες διαπραγματεύσεις ε, που θα καταλήξουν σε μια μακροχρόνια δέσμευσή μας στη χώρα και παρουσίασε ό,τι αφορά την αστυνομία του Αφγανιστάν μετά την εκπαίδευση που δίνουν η Ιούπολ και οι διάφορες ε, ε, χωροφυλακές, η Ιταλική και η Γαλλική εμπροκειμένου, βλέπουμε υψηλό βαθμό επαγγελματισμού ε, στην αστυνομία και εκτιμούν πάρα πολύ και η Αφγανοί και η διεθνής κοινότητα και όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί τη δική μας δράση, της Ιούπολ, ενώ στο παρελθόν δεν εκτιμούσαν πάρα πολύ την αστυνομία γιατί για λόγους που κατανοεί κανείς μέχρι τώρα ε, χρειαζόταν ε, παραστρατιωτική ε, ως αστυνομία, αλλά και περισσότερο η αστυνομία αυξάνει τη σημασία της και η εκπαίδευσή της θα πρέπει να μάθουν τι σημαίνει η αστυνόμευση της αστυνομίας πόλεων, ας πούμε, όπου να μην είναι στρατιωτική μονάδα ή παραστρατιωτική, που να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις γνώσεις. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων, αν έχει αλλάξει και πώς είναι η UPOL, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίως έχει αλλάξει. Πριν φτάσω, πριν από δύο χρόνια, οι Αφγανοί και η διεθνή κοινότητα ήταν σε σύγχυση ποιο εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα με γνωρίζουν οι συνάδελφοι, οι ε, συνομιλητές μου, έχουν και το κινητό μου τηλέφωνο. Θέλουν να μιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, ξέρουν ποιο να πάρουν. Έχουμε στα γραφεία μας ε, ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη και τα, 27, τα 17 που εκπροσωπούνται συνεργάζονται με τρόπο συνεκτικό για να επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν υπέρ της ασφάλειας και της ευημερία. και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Αυτά που ρώτησε ο κύριος Ζίγκερης για την κοινωνία των πολιτών και αν έχει γίνει πρόοδος τα τελευταία δέκα χρόνια ή τουλάχιστον τελευταία διετία που είμαι εγώ εκεί ναι, έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Να μοιραστώ μαζί σας. Πριν από μία διετία ε, εξεπλάγει πάρα πολύ και με έχει εντυπωσιάσει πόσο ζωντανή είναι η κοινωνία και πόσο έντονα και ελεύθερα είναι τα μίντια, τα μέσα ενημέρωση στο Αφγανιστάν. Είναι πολύ περισσότερο από άλλες χώρες που είναι στην άμεση γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, υπάρχει ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνίας των πολιτών. Είναι δύσκολη η λειτουργία τους, δεν έχουν χρήματα, δεν υπάρχει πλήρη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε και δεν επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις όσο θα ήθελα να είναι πραγματικά μεγάλη ανταμοιβή να βλέπεις περισσότερες γυναίκες στο κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνική και πολιτική ζωή του Αφγανιστάν. Νομίζω απάντησα για το μελλοντικό ρόλο της Γιούπολ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πακιστάν. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικός άμεσος γείτονα το Πακιστάν. Από τις επαφές που έχω εγώ και τις συνομιλίες με τους Πακιστανούς που έρχονται από το Ισλαμαμπάτ και από αλλού, διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει στάση ως προς τη δυναμική της περιοχής γενικά και το ρόλο του Αφγανιστάν ιδιαίτερα. Όπως είπε κάποιος, ο Πακιστανός, από την ηγεσία της χώρας. Είπε ότι θα ολοκληρωθεί η περιφέρεια και η συνεργασία εκεί όταν υπαστούν ε, το Αφγανιστάν στραφούν προς την Καμπούλ και παστούν του Πακιστάν προς την Ισλαμαμπάτ. Ε, οι δύο ηγέτες ε, των δύο χωρών επίσης προωθούν τη συμφιλίωση και πρόσφατα η Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν όταν ήρθε στην Καμπούλ όχι μόνο συνάντησε την κυβέρνηση αλλά τόνισε και το σεβασμό στην εδαφική ακαιρεότητα και τον πολυεθνικό χαρακτήρα του Αφγανιστάν. Συναντήθηκε με εκπροσώπους εθνοτικών ε, ομάδων, ε, Τατζίκους, Ουσμπέκους και άλλους ε, πολιτικούς ηγέτες της Βόρειας Συμμαχίας. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την προσοχή που δείχνετε για το Αφγανιστάν και θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή Εξωτερικών αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθούν περισσότερο με την ε, ε, τζίργα, την ε, συνέλευση την κοινοβουλευτική για να δημιουργηθεί και ένα πολυκομματικό πολιτικό τοπίο στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ουζάκας για αυτή την συζήτηση. Συμφωνούμε με τα όσα είπε ο κύριος Ζιγκέρης. Σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε εκεί. Και θα ειδωθούμε στο μέλλον πολύ περισσότερο λόγω των σημαντικών εξελίξεων που θα υπάρξουν και των ευθυνών που θα έχουμε μέχρι το 2014. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη.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 ε, καλωσορίζω την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, την κυρία Κλοντ Φων Αγνού. Η σημαντική οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Μα δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνεκμετάλλευση και ο επιμερισμός ε, στον αμυντικό τομέα ε, και οι ευκαιρίε που υπάρχουν για συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε? και μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ιδέες ε, και να μας σχολιάσετε την επερχόμενη συνοκορυφή κορυφή στο Σικάγο. Ε, δόθηκε μεγάλη προσοχή στις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο δυναμικού. Αυτό φαίνεται και από τις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει νομίζω να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έρευνα, στην βιομηχανία και στη συνεργασία στον ερευνητικό και μηχανικό τομέα, ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν θα έχουμε περισσότερα λεφτά, λιγότερα λεφτά ε, στο μέλλον. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Ε, υπάρχουν περιορισμοί και των αμυντικών προϋπολογισμών σε διάφορες χώρες. Ε, επομένως υπάρχουν και πιέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σε οικονομικό επίπεδο. Ε, ποια είναι η απόψή σα γι' αυτό τώρα που βρισκόμαστε στο, εν μέσω διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Αγνού, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να μιλήσω αγγλικά ή γαλλικά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μιλήσετε νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για σας να μιλήσω γαλλικά. Αλλά μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και να του πω ότι είναι μεγάλη τιμή που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σας. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε το διάλογο, συχνά συμμετέχω στο διάλογο στα πλαίσια της ε, υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Ο πρόεδρος υπενθύμησε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ε, είναι μια κρίσιμη στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα και μάλιστα όχι την ε, επιλογή, τη δυνατότητα, χάρη στη συνεργασία, χάρη στην κοινή προσπάθεια, χάρη στις συνέργειες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να έχουμε, αποκτήσουμε τα μέσα, ούτως ώστε η Ευρώπη να προασπίσει την ασφάλειά της. με τη χρησιμοποίηση των πολιτικών που έχει στη διάθεση της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε την πρωτοβουλία που ξεκίνησε για την εκμετάλλευση και τον επιμερισμό στη Γάνδη πάνω από ένα χρόνο, στα τέλη του 2010, ε, λίγο πριν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Μόναχο ξεκινήσει την ε, πρωτοβουλία για την ε, έξυπνη άμυνα είναι ουσιαστικά η ίδια προσέγγιση, ο ίδιος στόχος. Δηλαδή με προϋπολογισμούς πιο περιορισμένους, ανάλογα με το κράτος μέλος βέβαια, αλλά με, με προϋπολογισμούς ε, συρρυκνωμένους λόγω της οικονομικής κρίσης, παρόλα αυτά ε, να αναλάβουμε οι Ευρωπαίοι τις ε, ευθύνες μας για να υπρασπίσουμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας. Υπάρχει ένα δίλημα που πρέπει να επανεξετάσουμε και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε τα μέσα για να προωθήσουμε την ασφαλειά μας. Αυτή η εκμετάλλευση και επιμερισμό, το pooling και sharing δεν είναι μια ακόμα εναλλακτική λύση, αλλά μια κατεπίγουσα ανάγκη. Ε, ενισχύεται και από το στρατηγικό πλαίσιο και από το μήνυμα που περνάει από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ότι εσείς Ευρωπαίοι θα πρέπει να είσαστε πάροχοι ασφάλειας να συνεισφέρετε στην ασφάλεια και ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να προωθήσετε αυτή την προσπάθεια, να συνεισφέρετε κι εσείς στην εξασφάλιση της, του security της ασφάλειας. Η πρόοδο γίνεται ολοταχώ. Ε, στην στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα λάβαμε μία εντολή από του υπουργού να προωθήσουμε συγκεκριμένα project, σχέδια, ούτω ώστε να δείξουμε ότι αυτή η θέληση στην εκμετάλλευση και επιμερισμού, pooling και sharing, δεν είναι μια έννοια αφηρημένη, δεν είναι λόγια, δεν είναι μια απλή θέληση, αλλά μπορεί να γίνει και πράξη. Θέλαμε λοιπόν το συντομότερο δυνατόν και με βάση του εφικτού και με βάση του τι θέλουν να κάνουν διατηρώντας την κυριαρχία του στα κράτη-μέλη. Γιατί το δυναμικό είναι δυναμικό των κρατών μελών και οι αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση αυτού του δυναμικού είναι κυρίαρχες αποφάσεις των κρατών μελών, να δούμε πού είναι έτοιμοι να μοιραστούν και πού μπορούμε να προωθήσουμε και να προτείνουμε δράσεις ε, που να έχουν προστιθέμενη αξία. Ε, για το pooling και sharing. Προτείναμε λοιπόν δράσεις σε τομείς ε, όπου τα λεπτά θέματα της κυριαρχίας είναι λιγότερο ορατά και κυρίως της επιχειρησιακής ε, κυριαρχίας στα θέτρα των επιχειρήσεων. Γιατί είναι οι εθνικές διαδικασίες για την απόφαση ανάπτυξης στρατιωτικού εξοπλισμού, στρατιωτικών δυνάμενων. Ε, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαλειτουργικότητα και μια συνεργασία μεταξύ ε, Ευρωπαίων. Ό,τι είναι ε, εκπαίδευση, επιμελητεία, συντήρηση ε, και εκεί όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε σε θέατρα επιχειρήσεων όπου τα θέματα όπου δεν υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις, όπου είναι λιγότερο λεπτό το, το θέμα του αν θα πάνε ή όχι. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στην εκπαίδευση. Είχαμε ήδη προωθήσει δράσεις ε, για τον εξοπλισμό και, και το προσωπικό των ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης στο θαλάσσιο τομέα για την ε, ιατρική υποστήριξη, ε, νοσοκομεία εξτρατείας, δηλαδή, που είναι σημαντικά για την ασφάλεια των στρατιωτών μας όταν τους στέλνουμε σε θέατρα επιχειρήσεων και για τη θαλάσσια εποπτεία προωθήσαμε τέτοιε δράσει. Και κάτι που είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Εκεί που είμαστε ανάμεσα σε υποστήριξη και σε επιχείρηση, είναι το, η δράση για την, τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ε, κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ε, όλοι οι υπουργοί ήθελαν να προχωρήσουμε εκεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εντοπίσαμε τα χάσματα, τα κενά των Ευρωπαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε επιχειρησιακά με ικανοποιητικό τρόπο και όπου θα πρέπει και να έχουμε το δυναμικό και να υποφεληθούμε από το κοινό μας, ε, την κοινή μας προσπάθεια, στην κατάρτιση, στον ανεφοδιασμό κτλ. Ε, τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι είναι ένας τομέας όπου ρυθμίζουμε θέματα κυριαρχίας των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας αυτό το δυναμικό όταν το χρειαζόμαστε σε ένα θέατρο επιχειρήσεων. Πέρα από αυτές τις βραχυπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες δράσεις ε, ε, βάσει των οποίων ε, δεσμεύτηκαν η Υπουργεία. Όταν ε, συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια του άτυπου γεύματος με την Προεδρία της Λέδης Άστον, είδαμε ότι υπάρχει μια αλλαγή προσέγγισης μακροπρόθεσμα. μπορούμε να έχουμε σημαντικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά αυτή η προσπάθεια συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού ε, υλοποιείται μόνο μακροπρόθεσμα. Ε, αυτές οι εμπειρίες, ε, οι θετικές εμπειρίες στην εκμετάλλευση και του επιμερισμού είναι κυρίως ε, περιφερειακές. Στο Μπενελούξ, ε, στην ε, σκαρναδική συνεργασία, αλλά και σε διμερές επίπεδο είχαμε θετικά αποτελέσματα. Από αυτή την διμερή ή περιφερειακή συνεργασία Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε, τι μπορούμε να διδαχτούμε ε, από τις προσπάθειες άλλων ομάδων, δηλαδή, ούτως ώστε να το συνεχίσουμε και να το εφαρμόσουμε και εμείς στην περιοχή μας, στην ομάδα μας. Πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία και πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα της κυριαρχίας για να προωθήσουμε στην εκμετάλλευση για τον επιμερισμό. Επίσης, όταν κάνουμε οικονομίες σε ένα τομέα, πώς μπορούμε να ε, επανεπενδύσουμε αυτές τις οικονομίες. Παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος Μπρόκμι ανέφερε την έρευνα και την τεχνολογία. Αν δεν διατηρήσουμε α, τη δυνατότητα επενδύσεων στην έρευνα και στην τεχνολογία σήμερα, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο μη επιστροφής. μπορεί δηλαδή οι Ευρωπαίοι να μην έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν την τεχνολογική ανεξαρτησία ε, προς όφελος της ασφάλειάς τους. Μακροπρόθεσμα, αυτό που μας ζήτησαν οι υπουργοί την περασμένη εβδομάδα, με βάση ένα έγγραφο που ετοίμασαν τέσσερα κράτη-μέλη, το Βέλγιο, την Ελλάδα, η Φιλανδία και το Λουξεμβούργο ετοίμασαν αυτό το κείμενο, προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε μακρο, μακροπρόθεσμα τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που αναπτύσσονται στις ε, Βρυξέλλες και τη λογική που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μεταρρυθμίσουν και να ε, γράψουν στην, ε, όλες αυτές τις προσπάθειες στην εθνική, στον εθνικό τους σχεδιασμό. Και επίσης πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτή την πολιτική με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Τελευταίο σημαντικό στοιχείο και χαίρομαι πραγματικό που το σχολιάζω λίγο μετά το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ε, είναι το θέμα της συνεργασίας. Θέλω να δείξω στα κράτη-μέλη και να τα καθησυχάσω ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμπληρωματικό από αυτά, σε σχέση με αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν επικαλύψει. δεν γίνονται τα ίδια, υπάρχει συμπληρωματικότητα. Μιλάμε παραδοσιακά για ένα απόθεμα δυνάμεων. Ε, δεν ε, κάνουμε τα ίδια, αλλά θέλουμε να υπάρχει ε, συμπληρωματικότητα. Ο κύριος Ράσμουσεν μίλησε για τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στι επαφές μας με τον ΝΑΤΟ δείξαμε, δείξα, φάνηκε ότι αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Και <clears throat> φάνηκε ότι αυτή την έλλειψη που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Το δεύτερο παράδειγμα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι στον τομέα των ιατρικών, όπου τα κράτη-μέλη αποφάσισαν και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ να παίξουν το ρόλο τους, εξασφαλίζοντας ότι θα, οι προσπάθειε θα είναι συμπληρωματικέ. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δουλέψουμε ε, για τα, τη δυνατότητα ε, δημιουργίας νοσοκομείων εκστρατεία, συναρμολογούμενων. Και το ΝΑΤΟ ε, προσπαθεί να α, τυποποιήσει αυτά τα εξαρτήματα νοσοκομείων με βάση την εμπειρία που έχει από το Αφγανιστάν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας εξηγήσαμε τη συνεργασία που κάνουμε με τον ΝΑΤΟ. Ε, ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ήρθε και την περασμένη εβδομάδα με τον ε, στρατηγό Αμπριάλ ε, προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη για να σας αποδείξουμε ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα των προσπαθειών μας, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα μακροπρόθεσμα, πάντα για τους μακροπρόθεσμους στόχους, θέλουμε τα κράτη-μέλη να εντάξουν αυτή την προσέγγιση συνεργασίας στις, ε, στον εθνικό σχεδιασμό και στην εθνική μέθοδό τους και χωρίς να πω σε τεχνικά θέματα, θέλω να πω ότι τα εργαλεία που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας θέλουμε να ε, εξυπηρετήσουν και την εθνική προσπάθεια. Έχουμε ένα μηχανισμό ανάπτυξης ε, δυναμικού και θέλουμε αυτό το δυναμικό να χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να αναπτύξουν το, τη συνεργασία αυτή και τον επιμερισμό, την εκμετάλλευση και τον επιμερισμό. Δεύτερον, στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, στον EDA, ε, πρέπει να εντοπίζουμε τις ανάγκες των στρατιωτών μας, αυτή είναι το καθήκον μας. Επίσης, να δούμε τι προσφέρει η αγορά, η βιομήχανη για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Έπειτα, τι προσφέρει η έρευνα και η τεχνολογία ως λύσεις. Τι μπορεί να προσφέρει ε, αύριο μεθαύριο, ούτω ώστε να δούμε πώς όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε για να δούμε το δυναμικό που μπορούμε να αποκτήσουμε. Όλα αυτά είναι μοναδικά που κάνουμε. Ε, πουθενά άλλο δεν γίνεται αυτό, παρά μόνο σε εθνικό επίπεδο προφανώς, όπου μπορούμε την τεχνολογία και τη βιομηχανία, την έρευνα να τις δούμε από κοινού για να δούμε πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των στρατιωτών που αποστέλνουμε στα θέατρα των επιχειρήσεων. Η το άλλο επίπεδο ε, είναι ε, η, η, σχέση με τις άλλες ε, ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, πρόεδρε, αναφέρατε την ε, σχέση με την έρευνα. Προφανώς είναι σημείο κλειδί αυτό. Ούτως ώστε κάποιες τεχνολογίες, ξέρετε, ξέρετε κάποιες τεχνολογίες, κάποιες κάποιοι τομεί είναι ούτε στρατιωτικοί ούτε πολιτικοί. Ε, το διάστημα, α πούμε. Οι, συμπε... οι κυβερνοτεχνολογίες, η προσπάθεια καταπολέμησης των χημικών, ε, μικροβιολογικών, ε, πυρηνικών και ακτινολογικών όπλων, ας πούμε. Αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι ούτε στρατιωτικές ούτε πολιτικές αστικές. μαζί με τους υπόλοιπους ε, ευρωπαϊκούς φορείς προσπαθούμε να δούμε τις ε, συνέργειες με απόλυτο σεβασμό των ε, διαδικασιών που είσαστε θεματοφύλακες εσείς. Ε, στα πλαίσια του, της στρατηγικής Ευρώπη 2020 πάντα. Αναφερθήκατε στον προϋπολογισμό του οργανισμού μας. Φυσικά είναι γελίο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι 30 εκατομμύρια ευρώ είναι πολιτικό το θέμα. Ε, δεν είναι πολύ εύκολο να πει κανεί ότι εγώ θα αυξήσω τον προπολογισμό ενό οργανισμού στι Βρυξέλλε. Τουλάχιστον να μην μειωθεί όμω, ούτω ώστε να μπορέσει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα να κάνει αυτό που περιμένουν οι Υπουργοί Άμυνα. Αυτό που έχει σημασία πέρα από τον προπολογισμό και το μέγεθό του βέβαια είναι οι πιστώσει που μπορούν να δώσουν τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένα project που του ενδιαφέρουν ε, και όπου χρειάζονται επιπρόσθετες πιστώσει. Ε, Προ τα κονδύλια. Ε, έχουμε ακόμα 100, 150, 200 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώνουν τα κράτη-μέλη και προωθούνται χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση κάποια ερευνητικά προγράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, ε, με σεβασμό βεβαίω των διαδικασιών. Αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν χάρη στα δικά του στις δικέ του πιστώσει και στι πιστώσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό θέμα είναι ε, το Single European Sky, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, το πρόγραμμα CESAR ιδίως όπου προσπαθούμε όλες οι στρατιωτικές ανάγκες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον ένα αέριο έλεγχο, αλλά όλο το δυναμικό να λυθεί υπόψη, να εντοπιστεί και να λυθεί υπόψη. Και εμείς ως οργανισμός να είμαστε ο χώρος όπου τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους, τα εθνικά τους συμφέροντα. Και χάρη σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό ουρανό, οι στρατιωτικοί μπορούν να συνεχίσουν την αποστολή τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος, αλλά και να συνεισφέρουν θετικά με την αποστολή τους. Ελπίζουμε τώρα με τη δημιουργία της Task Force που οργανώνει η Κομισιόν να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια και χαιρόμαστε για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα πλαίσια αυτής της Task Force. Συμπερασματικά, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Μπορεί η, Ευρω... η Ευρώπη να να απολέσει ένα τμήμα του δυναμικού της για να εξασφαλίσει την ασφαλειά της. Γι' αυτό η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας είναι πολύ σημαντική για την προάσπιση των αξιών και των συμφερόντων μας. Επίσης, πρέπει να δείξουμε απέναντι στους εταίρους μας ότι παρέχουμε ασφάλεια, ότι είμαστε πάροχοι ασφάλειας, security providers. Αυτό το μήνυμα στο στις πολιτείες 38. Ε, είναι φυσικά πρόκληση, αλλά και είναι και ένα σημαντικό κίνητρο. Ποτέ δεν είχε εκφραστεί τόσο σαφώς να αποκτήσουμε το δυναμικό, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους εταίρους μας ανά τον κόσμο αυτή την ασφάλεια. Εμείς είμαστε ε, ένα εργαλείο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, στην υπηρεσία των κρατών μελών για να το πετύχουν αυτό αλλά θα πρέπει να μας χρησιμοποιήσετε στο 100% των δυνατοτήτων μας. Ε, χάρηκα που οι Υπουργοί Άμυνα ε, στην τελευταία συνάντηση έδειξαν την βούλησή τους με πολύ συγκεκριμένο, με πολύ απαιτητικό τρόπο να μας χρησιμοποιήσουν. Ε, πρέπει να μας δώσουν βέβαια και την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη. Ε, και είναι φυσικά και εσείς, ε, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αρνού, ο συνάδελφος Κάλλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάλλερ, συγγνώμη. Καλωσορίζω την ε, κυρία Αρνού στην Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην υποεπιτροπή μας, ε, εκτιμούμε πολύ την δουλειά που κάνετε. Αναφέρατε και την ε, σχετική έκθεση του συναδελφού Βίζεκ. Ε, βεβαίως η ε, παρέμβαση μπορεί να είναι λίγο πιο εντατική από αυτή που θα επιθυμούσαν ίσως τα κράτη-μέλη. Ε, οι πρωτοβουλίες για το pooling and sharing ποιε θα είναι και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει επιφέρει σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. 311 νέα προγράμματα παρουσιάστηκαν πέρσι μάλιστα από τα κράτη-μέλη και σήμερα συζητούμε μόλις τα 11 από αυτά. Τα υπόλοιπα 298 που πήγαν, τι έγινε. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος ε, ως προς αυτά. Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα. Τι έχει γίνει με αυτά τα υπόλοιπα projects ή τι θα γίνει. Και αν δεν έχουν προτιμηθεί, γιατί δεν έχουν προτιμηθεί. Τώρα, για τους ε, στόχους για το 2010 και για την ε, διεύρυνση του χρονοδιαγράμματος ε, επαόριστον. Μήπως έχετε δει κάποια κενά στις δυνατότητες που υπάρχουν ε, σε σχέση με αυτά που επιτεύθυνσαν τελικά. Και να αναφέρω και ένα παράδειγμα. Το αναφέρατε κι εσείς. Για... Το ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και μάλλον είναι λίγο προβληματικό το σημείο που ε, βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό από αέρος ε, των αεροσκαφών. Ε, υποθέτω ότι οι δυνατότητες που έχουμε ως προς αυτό το τομέα είναι πολύ δύσκολες. Ο Ράσμουσεν είπε, εντάξει, εμείς έχουμε λίγες, αλλά οι Αμερικανοί έχουν πολλές. ναι, αλλά πάλι οι Αμερικανοί μπορούν να μας πούνε, αυτά είναι δικά σας προβλήματα, είναι δική σας η κατάσταση, εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε αυτό. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον εφοδιασμό από αέρος, ε, αλλά προφανώς ε, είναι, δεν, είναι, δεν μιλάμε για διεύρυνση του στόλου, μιλάμε για την κατάσταση κάποιων παλιών ε, αεροσκαφών προφανώς. Αν όντω αυτή είναι η κατάσταση ε, για του ε, δύο μεγαλύτερου ε, δυνάμεις που παρεμβαίνουν σε αυτό το project, τότε εμείς που ούτω ή άλλω έχουμε μειωμένε δυνατότητες, ποια θέση έχουμε. Και επίσης, πώς θα κλείσουν αυτά τα κενά στις δυνατότητες που έχουμε. Και επίσης, μιλήσατε για τον ορίζοντα 2020, υπάρχει μια γνωμοδότηση από τη ΣΕΔΙ ως προς αυτό, και Νομίζω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να, κλείσουμε αυτά τα κενά γιατί μιλούμε για πολιτικά και στατοτικά προϊόντα για την ενίσχυση των αποστολών και όλα αυτά ήδη έχουν προβλεφθεί. Εσείς τι άποψη έχετε αν θα μπορούσατε να ευχηθείτε ας πούμε κάτι ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι που θα πρέπει να θέσουμε ως προς, τον, ως προς τις στρατιωτικές και τις πολιτικές δυνατότητες που έχουμε και πώς θα μπορούσαν αυτά να συμπεριληφθούν στον όριο του 2020 έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί και πρόοδος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. I think, uh, Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς η στρατιωτική συνεργασία σε ό,τι αφορά και τις ε, προμήθειες και την σύνδεση με την έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρωτόγονο στάδιο. Και συμμερίζομαι και τις ε, ανησυχίες που εξέφρασε ο κύριος ε, Γκάλερ σε ό,τι αφορά την έλλειψη πρόοδου Όντως ε, φοβούμε ότι έχει υπάρξει υπαναχώρεση σε ό,τι αφορά τις φιλοδοξίες που είχαμε θέσει στον ε, τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Και εσείς ίδια μιλήσατε επανειλημμένα για την κυριαρχία. Δεν είναι ένας ε, όρος που ακούμε πολύ συχνά στους υπόλοιπους τομείς τουλάχιστον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προφανώς υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ όσων θέλουν την διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, αλλά λένε ταυτόχρονα ότι ευχαρίστως θα επιμερίσουν και θα συνεκμεταλλευθούν τα στρατιωτικά τους, τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Κάπου κάποιος ψεύδεται. Θα μπορούσατε να μας πείτε συγκεκριμένα αν εσείς θεωρείτε ότι η αγγλογαλλική συμφωνία άμεν, άμυνας είναι ευλογία ή κατάρα για την ε, ανάπτυξη της ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, γιατί νομίζω ότι μας αποσπά τελικά από τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε και ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να στοχοθετήσουμε καλύτερα τις ε, δυνατότητες που έχουμε ώστε να ενισχύσουμε τις, ε, τους πόρους και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την Τουρκία. Ποιο είναι το κόστος της μη συμμετοχής της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, αν και εγώ έχω έτσι μια διαφορετική οπτική, ε, το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Μιλήσατε και συγκρίνατε μάλιστα την, ε, τις διεθνείς προσπάθειες ε, για την δημιουργία, ας πούμε, ενός ε, νοσοκομείο για, με την, ε, και τη συγκρίνεται με, τη με, την, ε, με τις ιδιωτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και κάποιοι λόγοι για το γιατί τελικά η διαφάνεια και η εθνική κυριαρχία την χάνουν τόσο ευαίσθητης διαχείρισης ό,τι αφορά την εμπλοκή τους στους στρατιωτικούς τομείς. Εμείς Έχουμε ε, στην ε, Γερμανία συζητήσει ενδελεχώς το θέμα αυτό τη συμμετοχή σε ε, ένοπλες σειράξεις και γι' αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Τελικά, πώς λαμβάνετε υπόψη το ότι αυτό το κοινοβούλιο έχει κάποιες επιφυλάξεις. Μπορείτε εσείς να μας διαβεβαιώσετε ότι οι, αυτές οι κοινέ δυνατότητες μέσω της συμμετοχής, ας πούμε, και των γερμανικών ε, δυνατοτήτων των στρατιωτικών δεν θα επηρεαστούν αν ας πούμε το γερμανικό α, κοινοβούλιο αρνηθεί να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα pooling and sharing. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας πείτε εσείς πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό τελικά στην πράξη, αν κάποιο κοινοβούλιο αρνηθεί να συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια του pooling and sharing των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Άκουσα σωστά το όνομά μου κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριος Κύριλοφ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε ενώπιον μας. Έχω μια ερώτηση που έχει σχέση με το σχέδιο για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς που είπατε στο τέλος και πιο συγκεκριμένα Βεβαίω κατανοώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με προστιθέμενη αξία, αλλά έχει και κάποιες επιπτώσεις. Δεν μιλώ για το κόστο εδώ, για τις αεροπορικέ εταιρείε, που είναι μάλλον ίσον ζήτημα, αλλά σε ό,τι αφορά την πολεμική αεροπορία των διαφόρων κρατών, αυτό οπωσδήποτε θα επιφέρει, πώς να το πω, κάποιο σοβαρό επιπλέον φόρτο για τις απαιτήσει ενώ σε ό,τι αφορά κάποια μικρότερα κράτη-μέλη. Και μπορεί όλοι να ενδιαφερόμαστε ε, να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα πρέπει ε, σε ένα πρώτο στάδιο να βασιστούμε σε εθελοντική συνεισφορά από τον αμυντικό προϋπολογισμό της κάθε χώρας. Έχετε κάνει καμία μελέτη για τον υπολογισμό για το ποιο θα είναι το ειδικό βάρος ή το βάρος που θα πρέπει να σηκώσει το κάθε κράτος μέλος από πλευράς οικονομικής εκεί. Και αν υπάρχει τρόπος να κινητροδοτηθούν ορισμένες χώρες που μπορεί να έχουν ασύμετρες ε, οικονομικές επιβαρύνσεις για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Λίζεκ. Θα ήθελα ε, να πω ότι με την κυρία Αρνό έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες στη συζήτηση για τις ε, οικονομικές επιπτώσεις ε, της χρηματοοικονομικής κρίσης στον τομέα της άμυνας. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ήταν ε, ε, πολύ πολύτιμες οι συζητήσεις μας για την εκπόνηση της έκθεσής μου. Έχω δύο ερωτήσεις, μία γενικότερη και μία ειδικότερη. Θα αρχίσω από την ειδικότερη, είναι πιο σύντομη. Κυρία Αρνού, εσείς είστε ικανοποιημένοι προσωπικά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας από τη συνεργασία σας με τα κράτη-μέλη. Γιατί γνωρίζω ότι δίστανται οι απόψεις για τη συνεργασία και τη δέσμευση των κρατών μελών στα διάφορα έργα. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα. Είστε ικανοποιημένοι ε, από το ε, βαθμό και το επίπεδο συνεργασίας των νέων κρατών μελών. Και ένα δεύτερο, γενικότερο ερώτημα. Ας ονειρευτούμε λίγο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που θα θέλατε, ποιος θα ήταν ο ιδανικός ε, προϋπολογισμός για σας, για τον οργανισμό, για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε πλήρως στην αποστολή σας. Ευχαριστώ. I would like to thank you very much Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και για αυτό που μου είπατε να σας πω για τα όνειρά μου και να εκφράσω τις επιθυμίες και τις ευχές μου. Ε, αρχίζω από τις ερωτήσεις του κυρίου Γκάλερ. Τι έγινε με τις δυνατότητες 3 εν, 11. Ε, Α, ρωτήσατε τι έγινε για τα 3, 11, 11 τελικά και ποιες ευκαιρίες έχουμε. Θελήσαμε να δείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε άμεση δράση κατανοώντας και συμπεριλαμβάνοντας τη δράση μας ε, την πολύ δινή θέση στην οποία βρίσκονται τα κράτη-μέλη μας ε, τα οποία γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, που μπορεί να μην είναι δραματική η κατάσταση σε όλες τις χώρες, ε, αλλά είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και δεν ήταν πρόθυμα να επιλέξουν τα 300 έργα. Το ίδιο είναι και με το ΝΑΤΟ. Είναι 11 τελικά, αλλά με διάφορα στοιχεία. Αν δείτε τον εφοδιασμό στον αέρα είναι μία δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορα στοιχεία. Και μετά μπορείτε να ε, ενώσετε τους τομείς ή να τους ε, κατακαιρματίσετε για να βγάλετε διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Αλλά θελήσαμε να δούμε τι είναι όριμο, τι είναι έτοιμο να εφαρμοστεί και τι είναι εφικτό. Αλλά τα υπόλοιπα έργα δεν σημαίνει ότι τα ξεχάσαμε. Ούτε θέλουμε να τα ξεχάσει κανένας άλλος. Ένας πολύ σημαντικός τομέας έχει να κάνει με την αερομεταφορά και τα μαϊταγωγικά αεροπλάνα. Όλα αυτά συνεχίζονται και μπορεί να μείνει σε πολύ ορατό επίπεδο. Ε, και μάλιστα το συζήτησαν και οι υπουργοί. Θα πρέπει τους στόχους να τους προβάλλουμε, να τους διαφημίζουμε ή να είναι πολύ χαμηλή η πτήση και να ξεφεύγει και από τα ραντάρ, να μην την παίρνει είδηση κανείς. Αυτό έχει να κάνει με τα κράτη-μέλη. Ως εκτελεστική διευθύντρια και εγώ στον οργανισμό ε, είμαι... Ε, υποχρεωμένη να υποστηρίζω τα κράτη ανάλογα με την πολιτική τους ε, επιλογή και να βοηθούμε όσοι μπορούμε. Ε, όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Εμείς αναφέρουμε, κάνουμε προτάσεις στους υπουργού σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ας πούμε, για τα αναγνωριστικά, ας πούμε, δεν έχει καλυφθεί, είναι ένα ευρύ πεδίο, αλλά έχει ε, αντιμετωπιστεί σε πολύ μικρό βαθμό από τους Υπουργούς Αμήνης και επανειλημμένα θα ερχόμαστε με νέες προτάσεις. Το ίδιο έχει να κάνει με μελλοντική ε, παρατήρηση και επικοινωνία μέσω δορυφόρων. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε αυτό και περαιτέρω όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διάστημα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό σε ό,τι αφορά το διάστημα, ε, είναι πραγματικά ε, ένας κλάδος που κατεξοχήν θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα έδειξαν πόση σημασία έχει να εργάζεται κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ορίζοντα 2020 που μου είπατε να κάνω μια ευχή ποιο θα ήταν το ιδεώδες πεδίο εργασίας προσωπικά ως άνθρωπος είχα την τάση να κάνω ένα μακρύ ευκολόγιο. Σας είπα την κυβερνοτεχνολογία, CBRN, ε, τις ναυτικές επιχειρήσεις. Ε, αν θέλετε, αν ε, μου επιτρέπετε να επικεντρωθώ σε κάτι που έχουμε εργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τα τηλεκατευθυνόμενα συστήματα. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι εκεί και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Το drone, δεν ξέρω πώς ε, είναι στα αγγλικά. Ε, αλλά είναι διάφορα τηλεκατευθυνόμενα ε, σκάφη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς σκοπούς, όχι μόνο για στρατιωτικούς, με διαφορετικό εξοπλισμό κάθε φορά. Αυτό που κάνουμε εμείς στον οργανισμό μας είναι ότι έχει να κάνει με επιστοποίηση, με ε, κανονισμός με διαλειτουργικότητα των ε, στοιχείων αυτών για να μπουν ε, σε ένα αέριο χώρο που δεν είναι διαχωρισμένος θα πρέπει να έχουν και την απαραίτητη τεχνολογία για να μπορούν να πετούν με ασφάλεια σε κάποιο αέριο χώρο και των πολιτικών αποστολών. Είναι δαπανηρό να αναπτύσσονται αυτά τα προγράμματα και αυτά τα στοιχεία και είχαμε μία επίδειξη που ήταν πάρα πολύ δαπανηρή στον οργανισμό μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συγκλίνουν και οι πόροι και να έχουμε κοινού στόχους, και ο κοινοτικός προπολογισμό και ο προπολογισμό του κάθε κράτους μέλους. Και αν μου επιτρέψετε να πω και μια τελευταία ευχή, εκεί να επικεντρωθούμε, γιατί έτσι ε, αυτό είναι απόδειξη ότι οι δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ε, πολιτικούς σκοπούς και για στρατιωτικούς. Και είναι ε, σημαντικό αυτό και το θέμα της πιστοποίησης και ε, της ρύθμισης κάποιων κανόνων δηλαδή. Τώρα, ο νεφοδιασμός καυσίμου στον αέρα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έχετε δίκιο πραγματικά αν ή αν αυξήσουμε σημαντικά τις δυνατότητές μας, Υπάρχει υπάρξει μεγάλη διαφορά. Και ο καλύτερος τρόπος είναι οι κρατικές προμήθειες. Αλλά υπάρχει διαφορετικός τρόπος κάθε φορά να γίνει. Ε, μπορεί κάποιος να αγοράσει αεροσκάφη, ας πούμε, για να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι εξασφαλίζει ότι έχει τις δυνατότητες και ότι δημιουργείται και ένας σύνδεσμος με την αμυντική ε, βιομηχανία, στην EDTIB, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Βάση. Αλλά δεν είναι μόνο αγορά σε αεροσκάφη. Ε, σε κανονικούς καιρούς ε, έχουν τα κράτη-μέλη πλεόνασμα στι ώρες πτήσης. Αλλά εμείς θέλουμε τα κρατημέρη να αποκτούν εξοπλισμό, αλλά με τον ίδιο αριθμό αεροσκαφών, εάν ε, συνδυάσουν, ε, έχουν συνεκμετάλλευση και για τις ώρες πτήσης και για την εκπαίδευση ε, και για τα τεχνικά και τον εξοπλισμό, έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τις πλεονάζουσες δυνατότητες που έχουμε εφόσον έχουμε εξορθολογήσει την υποστήριξη. Κύριε Ντάφ, εγώ δεν μπορώ να σας πω εάν συμφωνώ ή όχι. Εάν συμμερίζομαι την απογοήτευσή σας, δεν είναι δική μου δουλειά να το πω αυτό. Αν μπορώ παρόλα αυτά να εξηγήσω γιατί μίλησα για την έννοια της κυριαρχίας, ε, είπα κατ' επανάληψη αυτή τη λέξη, ε, ειδικά όταν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Ε, δεν το χρησιμοποιούμε την ίδια συχνότητα όπως τον όρο νόμισμα, ας πούμε. Ε, τώρα έχουμε το, την Ευρωζώνη και το Ευρωπαϊκό Νόμισμα. Αλλά στο τομέα της άμυνας, ε, ακούστηκε, υπάρχει το θέμα του τι θα πούν τα εθνικά κοινοβούλια. Το ερώτημα αυτό το, ακούσαμε και από ευρωβουλευτέ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το σεβαστούμε. Είναι μια πραγματικότητα. Ε, σε, στα κράτη-μέλη έχουμε κάποιε πολιτικέ διαδικασίε με βάση τι οποίε αποφασίζεται εάν το κράτο μέλο εμπλέκεται σε μια διένεξη ε, και αν θα αναπτύξει στρατιωτικό δυναμικό. Είναι θέμα κυριαρχία. Και το στατιωτικό δυναμικό που έχει κανείς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την ΕΠΑ, ας πούμε. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για εθνικούς σκοπούς, για επιχειρήσεις ανατοικές ή για επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Αυτό ονομάζω κυριαρχία. Και για να απαντήσω το ερώτημα για την Bundestag. Εμείς ως οργανισμός θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα διαφορετικά συνταγματικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για να αποφασιστεί. Το κάθε κράτος μέλος αποφασίζει από μόνο του αν θα αναπτύξει το δυναμικό του και εμείς πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε σε δύο πράγματα. Το ένα το ανέφερα ήδη, είναι οτιδήποτε δεν έχει να κάνει, ότι δεν είναι ό,τι αφορά την συντήρηση, την επιμελητία κτλ. Θέματα που δεν είναι ευαίσθητα σε σχέση με την κυριαρχία όσο περισσότερο μοιράζεσαι πράγματα, τόσο θα πας προς κάτι που είναι ευρωπαϊκό. Και όμως αυτά τα θέματα είναι πιο αποδεκτά. Δεύτερο είναι να λάβουμε υπόψη τις θετικές εμπειρίες που είχαμε και τις θετικές διατάξεις και ό,τι θετικό προέκυψε από κάποιες πρωτοβουλίες. αν πάρετε, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Διοίκηση α, Εναέριας Μεταφοράς, ε, χρησιμοποιήθηκε στην Λιβύη Ορισμένα κράτη-μέλη έκαναν αυτό που τους επιτρεπόταν πολιτικά και που χωρίς να τους δημιουργεί πρόβλημα. Για την αγγλογαλλική συνθήκη. Έχω Σκοτσέους συνεργάτες κάθε μέρα κάθε μέρα συνεργάζομαι με αυτούς και θα μιλάγα για βρετανογαλλική συνθήκη. Δεν μπορώ να μιλάω για, δεν είναι σωστό να μιλάω, πολιτικά ορθό να μιλάω για αγγλογαλλική συνθήκη. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφεληθούμε από αυτήν. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή μας. Καταρχάς δείχνει το επίπεδο εμπιστοσύνη. που μπορεί να κυριαρχεί ανάμεσα σε δύο κράτη-μέλη. Ε, δύο κράτη-μέλη τα οποία έτσι, από τη φύση τους έχουν και κάποια, κάποιο βαθμό δυσπιστίας το ένα, το ένα απέναντι στο άλλο. Όταν πολιτικά όμως επιθυμείς ένα επίπεδο εμπιστοσύνης, το οικοδομείς. Και αυτό συνδέεται με το θέμα της ε, κυριαρχίας. Τότε υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, ούτως ώστε να εξασφαλίσεις αυτή την ε, εμπιστοσύνη με σεβασμό των εθνικών διατάξεων. Κάποιες ε, διατάξεις έχουν αναπτυχθεί σε αυτά πλαίσια αυτής της Βρετανογαλλικής ε, συμφωνίας που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Και για την Ορντευκό και για την συνεργασία Benelux, δηλαδή και για τη σκανδιναμική συνεργασία και για τη συνεργασία Benelux. Μπορούμε να το κάνουμε. Στη, στην EDA ε, προτείναμε ορισμένα πράγματα για την ε, θαλάσσια συνεργασία. Ε, τα προτείναμε στη Γαλλία και στην ε, Βρετανία. Και εμείς ως EDA α, εποπτευουμε ούτως ώστε όταν θελήσουν κάποια κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία μπορέσουν να το κάνουν. Για το ΣΕΖΑ Πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να προβλέψουμε όλα τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το τελικό κόστος. Το τελικό κόστος ε, το αποτιμούμε στα 7 δις. Ε, συχνά συζητώ μαζί σας το θέμα του ΣΕΖΑΡ. Αυτό το νούμερο θα πρέπει να το ξαναδούμε, θα πρέπει να χτενίσουμε τους υπολογισμούς. Ε, γιατί μπορεί τελικά να καταλήξουμε σε ένα ποσό πολύ διαφορετικό από τα 7 δί. Θα πρέπει να μπούμε στι λεπτομέρειες και του πόσο θα κοστίσει το κάθε είδους ε, στοιχείο του capability του δυναμικού. Και όταν βάζεις και νέα στοιχεία θα πρέπει να ξαναπηγαίνεις και να ξαναβλέπεις την οικονομική αποτίμηση, το πόσο κοστίζει. και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προλάβουν τις απαιτήσει ε, για το ΣΕΖΑΡ και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα πράγματα. Εμεί θέλουμε οι ανάγκε των κρατών μελών να ληφθούν υπόψη, οι εθνικέ ανάγκε. Και όλη η δουλειά που γίνεται στο Eurocontrol για το ATM. καθώς και οι ειδικέ ανάγκες του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Επίσης ξέρετε ότι η Κομισιόν προτείνει να δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ, 3 δις ευρώ, συγγνώμη, που δεν θα, μπουν, δεν θα πάνε κατευθείαν σε στρατιωτικούς φορείς, αλλά επαναλαμβάνω, κάποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά και πολιτικά. Τελευταίο στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ τον τελευταίο μιλητή και σας ευχαριστώ για την προσφερόμενη συνεργασία και την συνεργασία που θα έχουμε όταν ετοιμάζετε την εκθεσή σας. Η αξιολόγηση της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Πάντα θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, το πλήρες δυναμικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Γι' αυτό προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε δράσεις ε, συχνά κάνουμε κάποια πράγματα έτσι πολύ μυστικά και ταπεινά θα έλεγα, που δεν τα ξέρουν οι υπουργοί. Ε, κάποια άλλα προγράμματα όμως τα κάνουμε ε, και τα ξέρουν πολύ περισσότερο. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα παλιά χρησιμοποιούν περισσότερο τον οργανισμό και τα καινούργια λιγότερο. Δεν, υπάρχει, δεν είναι εκεί η διαφοροποίηση. Τώρα, ο ιδανικός προπολογισμό εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε μια υπηρεσία προμηθειών, το οποίο νομικά είναι δυνατόν. Αλλά θέλουμε, πρέπει να δούμε αν το θέλουν τα κράτη-μέλη. Ε, αν βάλουμε ακόμα ένα μηδενικό, ε, δεν φτάνουμε στα 30, φτάνουμε στα 300. 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάποια στιγμή τα κράτη-μέλη θεωρήσουν, πιστέψουν ότι θέλουν περισσότερα πράγματα τότε μπορούμε να ασχοληθούμε και με τις προμήθειες και να αναπτύξουμε και μια μέθοδο για τις προμήθειες. Αλλά δεν θέλω να βάλω ένα ποσό εκεί ότι θέλουμε ένα ακόμα μηδενικό, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε αύξηση 2%. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν, δεν παίζεται έτσι ο προπολογισμό. Θέλουμε να δούμε σε τι αποστολέ θα, θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη ότι είναι χρήσιμε για τον EDA, για τον οργανισμό μα. Και ο προπολογισμό πρέπει να ακολουθήσει. Προ το παρόν, πρέπει απλώ να είμαστε μια βιώσιμη υπηρεσία, ένα βιώσιμο οργανισμό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένα σχέδια. Αυτό, αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγνού. Κάποια στιγμή έφυγα από την αίθουσα. Uh, Το συγγνώμη. Αλλά σας είπα από την αρχή. Το θέμα των ε, συρρυκνωμένων προϋπολογισμών υπάρχει παντού. το θέμα της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό πρέπει να το συζητήσουμε. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός που έχει ειδικό καθεστώς. Υπάρχει ένας πιο έντονος περιορισμός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό το προσωπικό μας ανανεώνεται έντονα. Έχουμε εμπειρογνώμονες που κάθονται για λίγο, αποσπόμενοι από τα κράτη-μέλη. Ε, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε την επαφή με τα κράτη-μέλη, γι' αυτό έχουμε αυτές τους αποσπόμενους. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα λοιπόν σε σχέση με το προσωπικό που έχουμε και άρα και με τον προπολογισμό. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η σχέση με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικά είναι δυνατό να συνδεθούν οι δύο προπολογισμοί. Μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι για τη χρηματοδότηση του προσωπικού, αλλά για χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων. Εσείς πρέπει να το αποφασίσετε πολιτικά απλώς ε, το θέλετε. Αλλά νομικά μπορεί να γίνει αν το θέλει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ και φοβόμουν αυτή την απάντηση. Σας απογοήτευσα δηλαδή. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα, να το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Wir müssen jetzt schnell machen. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τρέξουμε. Για τον προπολογισμό δεν θα προκάνουμε, γιατί αρχίσαμε δυόμιση και σχολάμε σε λίγο. Ε, λόγω των κανόνων μας θα πρέπει να κλείσουμε στις 6 και επειδή πρέπει να ψηφίσουμε, παρακαλώ σύντομα όμως να συζητήσουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Παλέτσκης, να μας κάνει μια σύντομη ε, παρουσίαση και αν χρειάζεται να μας ενημερώσει για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. επίζω να σας άρεσε η συνεδρίασή μας και θα παραμείνουμε σε επαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τη συνεργασία στον τομέα της ε, ενεργειακής πολιτικής και τους, με, τους, με τους πέραν των σύνορων μας Υπάρχει μια έκθεση η οποία εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε μάλλον από το Κοινοβούλιο πριν από πέντε χρόνια. Ο κύριος Άρους Βόλσκι ήταν ιδιαίτερο ενεργός στο να υποβάλει ε, σημαντικές τροπολογίες. Τον ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπου βεβαίω συναδέλφους που υπέβαλαν συνολικά 44 τροπολογίε. Οι περισσότερες έχουν γίνει αποδεκτές από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Το έγγραφο αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ευρεία συνένεση για την ανάγκη ύπαρξης ενεργειακής πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και, σε επίπεδο, ε, αλλά και με τους εταίρους μας πέραν των συνόρων μας. Προφανώ, ε, ε, κάποιε από τι τροπολογίε εμπίπτουν στην ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή που είναι η Ήτρα, η οποία επίση εκπονεί τώρα μια έκθεση για τους... υπάρχουν έξι συμβαστικέ τροπολογίε από του Κιώδη. Υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία τα οποία τονίζονται στην έκθεση. Καταρχάς, λόγω της ε, μεγάλης εξάρτησης της, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εισαγωγέ ενέργειας και των προβλημάτων που υπάρχουν για την ε, διαμετακόμιση της ενέργειας, Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τονίζουμε ότι ε, οι, ενεργειακές σχέσεις θα πρέπει να ε, συμβάλλουν για την προώθηση των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θε, θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία, υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων κτλ. Άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι ότι πρέπει να υπάρξει στενότερο συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, έτσι ώστε να μπορούν να δρουν από κοινού σε θέματα που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια. Άλλο ένα σημαντικό σημείο, ειδικότερα σχετικό με τις ε, νέες χώρες, ε, ζητούμε από την Κομισιόν να, να παρακολουθεί και να μας ενημερώσει ε, για τα υψηλότατα πρότυπα που υπάρχουν στις χώρες που γυρνιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε από τις όμορες χώρες να να κάνουν στρες test στους που έχουν και στα εργοστάσια ενέργειας που έχουν. Ο κύριος Έρους Βόλσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο αρχίζαμε, αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε, όπως είπε ο κύριος Παλένσκης, πριν από πέντε χρόνια. να συγχαρώ τον κύριο Παλένσκη για το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε. Να ξεκινήσω όμως λέγοντας, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο, όχι επί της ουσίας, αλλά για το ότι η Επιτροπή μας έχασε την αρμοδιότητα που έχει στον τομέα αυτό της ενεργειακής πολιτικής και την καθήλυνα αρμοδιότητα πια την έχει η Ήτρε, σύμφωνα με τον κανόνα 50. Η Ήτρε λοιπόν είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και θα ζητούσα από τον Πρόεδρο να ε, με κάποιο τρόπο να ανακτήσουμε την αρμοδιότητα αυτή για τον τομέα τουλάχιστον της ενεργειακής πολιτικής στο μέλλον για να μην χάσουμε την ε, παράδοση που έχουμε, την κληρονομιά όλων όσων έχουμε κάνει ε, αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Το τελικό κείμενο νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Και όπως είπα, συγχαίρω τον κύριο Παλένσκης για το γενικό αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε. Επιμένουμε στον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, ε, διεθνή σκακέρα της ενεργειακής πολιτικής. Ζητούμε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Ε, θέλουμε επίσης και οι αντιπροσωπείες επιτόπου να ε, συμμετέχουν, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το ρόλο που έχουν να παίξουν. Ε, υπάρχει βεβαίως και η ανακοίνωση ώστε να παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την εξέλιξη των πραγμάτων στον τομέα αυτό τη ενεργειακή πολιτική. Να αναφερθώ τώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο τη έκθεση. Υπάρχει μια πολύ καλή συμβαστική πρόταση για τη Ρωσία, η νούμερο 4, και ζητώ από όλε τι πολιτικέ ομάδε να την υποστηρίξουν. Μια που είμαστε στα πλαίσια του κανόνα 50, θα ψηφιστεί η ογνωμοδότηση στην Λομέλεια και βεβαίω εγώ την υποστηρίζω ένθερμα. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Παλένσκι, του ε, Σκιώδη και όλου του υπόλοιπου συζητητέ για το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι από ό,τι φαίνεται. Να πω λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση. Ούτως ή άλλως έχει υποβληθεί το σχετικό κείμενο και από τον Επίτροπο Ετινιέρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περιβαλλοντική πολιτική. Όντω, ε, δυνάμει του κανόνα 50 η καθήλυνα αρμοδιότητα πήγε στην Επιτροπή Ήτρε. Και βεβαίω ε, ούτω ή άλλω ο ε, Επίτροπο Έτιγκερ είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι ο υπεύθυνο ο Επίτροπο Περιβάλλοντο. Οπότε ας μην παρεκκλίνουμε του στόχου μας. Υπάρχει κάποιος ε, αρμόδιος υπουργός ε, για το θέμα αυτό. Για να έχουμε λοιπόν και την ε, απαραίτητη τάξη. Ας δούμε τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες των επιτροπών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο γιατί εν τω μεταξύ, όπως έχει πει και η διάσκεψη των Προέδρων, υπάρχει τέτοιος αγώνας, γίνεται τέτοια μάχη για τις ε, ε, αρμοδιότητες που στο τέλος θα χάσουμε 4-5 μήνες για να μπορέσουμε να ε, μοιράσουμε τις αρμοδιότητες, οπότε χρησιμοποίησαμε αυτό το άρθρο 50 για να γίνει αυτή η κατανομή. Ε, τώρα αν σε κάθε ένα project που προκύπτει ή σε, κάποιο, σε οποιαδήποτε γνωμοδότηση που προκύπτει ε, αρχίζουμε να ζητούμε κατανομή αρμοδιοτήτων, θα τεθούν και οι στόχοι μας ένα αμφιβόλο. Ας στηρίσουμε λοιπόν τον ιστορικό κανονισμό που έχουμε ψηφίσει Τέσσερις, μόνο, τέσσερις μήνες ε, δεν έχουμε δραστηριοποιηθεί. Αυτό πραγματικά είναι τελείως παράλογο. Έχουμε ε, κανόνες ε, τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε. Και πρέπει βεβαίως και εμείς άμεσα να αρχίσουμε να δραστηριοποιηθούμε και πάλι. Για την άκρη του κυρίου Παλένσκης υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, σχόλια. Όχι. Οπότε αύριο θα την ψηφίσουμε. Α, η Κομισιόν μήπως θέλει κάτι να πει. Ευχαριστώ. Να πω απλώς ότι η Κομισιόν είναι ιδιαίτερως ικανοποιημένη και από την έκθεση και από τις τροπολογίες που υπήρξαν. Υπάρχει ήδη μια ανακοίνωση Κομισιόν από το Σεπτέμβριο και ήθελα να πω ότι η γνωμοδότηση όντω τονίζει την σημασία που έχει η ενεργειακή πολιτική για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τονίζει την ανάγκη που υπάρχει για ενισχυμένο συντονισμό και βεβαίω τονίζει και τι ενεργειακέ συμφωνίε που υπάρχουν ε, με τι τρίτε χώρε. Θέλω απλώ εδώ να αναφέρω κάποια πράγματα υπό το φω των ε, τροπολογιών που έχουν υποβληθεί σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, ε, οδικό χάρτη, η Κομισιόν έχει εκδώσει μια ανακοίνωση ε, όπου δεν υπογραμμίζεται μόνο οι προτεραιότητες, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος κατάλογος δράσεων που ορίζουν σαφείς δραστηριότητες που εφαρμόζονται, που βρίσκονται εν εξελίξη από τον Σεπτέμβριο. Οπότε η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα, ας πούμε τη συμφωνία με την Ρωσία και τη Λευκορωσία για τη διαχείριση των, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει η εντολή που έχουμε λάβει από τις αρχές του έτους, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις τον προηγούμενο μήνα. Δεύτερον, είναι σαφέ ότι η διμερεί και οι πολυμερεί συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφή ε, σημαντικό μηχανισμό για να εξασφαλίσουμε την ισότητα των ε, όπλων, την διαφάνεια ε, και την ισορροπία μεταξύ των σχέσεών μα και αυτό ισχύει για όλε τι για όλες τις συμφωνίε, όχι μόνο για τι εταιρικέ σχέσει. Και όταν μιλούμε για συμφωνία με τρίτε χώρε, πάντα προσπαθούμε να προωθούμε αυτέ τι αρχέ και τις σχετικές βεβαίως πτυχές του κοινοτικού κεκτημένου. Η αγορά μας είναι ανοιχτή σε συμμετοχή, τρίτων, σε συμμετοχή εταιριών από τρίτες χώρες. Επίσης δεν έχουμε συγκεκριμένες ρήτρε ε, στις συγκεκριμένες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε γενικές ρήτρε ε, ασφαλιστικές δικλείδες για τον ε, μηχανισμό έγκυρους προειδοποίησης που είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε περίπτωση τώρα μονομερών αλλαγών στις συμβάσεις αυτές, οι εταιρείες βεβαίως ε, πρέπει να ε, ε, εμπλακούν στις διαδικασίες διαιτησίας όπως προβλέπεται. Και επίσης η Αναγέννηση Κομισιόν ζητά να υπάρξει η δυνατότητα εκπόνησης μεγαλύτερων projects ενεργειακών με τρίτες χώρες Βεβαίω ε, εκεί υπάρχουν κάποιε ε, ρυθμιστικές και νομικέ ε, αβεβαιότητε, συνέπειε, οι οποίε καλύτερα την χάνουν διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει α πούμε στην περίπτωση τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Αζερβαϊτζάν και Τουρκμενιστάν για τον αγωγό από την Κασπία. Και πρέπει να πω ότι οι Αυτέ οι συμφωνίε δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές ή τον όγκο Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρης Βάσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το σχολείο σας, το σχολείο μου. Αλλά για να είμαστε σαφείς, Κατανοώ ότι το θέμα της ασφάλειας, της ενέργειας και της εξωτερικής πτυχής έχει λάβει ιδιαίτερη σημασία από τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ε, λέγοντας ότι είναι δική μας ε, αρμοδιότητα. Δεν ε, παρεμβαίνω εγώ στα χωράφια διαχωρισμών αρμοδιοτήτων μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου, αλλά τουλάχιστον δεν θα πρέπει και να μας υποδεικνύουν και σε εμά ποια είναι η αρμοδία επιτροπή που θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Εδώ δεν μιλούμε για ενεργειακό μείγμα, ούτε για πρόβλημα ενέργειας ε, ή βιομηχανικής, ε, ή ε, για πρόβλημα πολιτικής. Είναι θέμα ασφάλειας και αυτό έγινε αποδεκτό από όλη την Επιτροπή μας, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, οπότε θα πρέπει και εμείς να το δούμε ανεξάρτητα αν είναι στα χέρια της, ε, του Επιτρόπου Ενέργειας που κάνει μια εξαιρετική δουλειά ή αν ε, την χάνει διαχείριση αλλού ή από κοινού σε κάποιες επιτροπές. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά έκανες και το είπες. Που είπες ότι καμιά φορά για αυτά τα θέματα μπορεί και γερμανός πολιτικός να πει κάτι σωστό. Κάνουμε βήματα ένας προς την κατεύθυνση του άλλου. Εντάξει, αστείωμενο. Αυτά με τι αρμοδιότητες να τα πείτε με τον κύριο Αλμπερτίνη, γιατί εγώ τότε δεν ήμουν πρόεδρος. Το είπαμε. Δεν ξέρω κύριε Παλέτσικη, θέλετε να πείτε τίποτα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού θα μπορέσουμε να περάσουμε και πολλά πράγματα. Αλλιώς ήταν το άρθρο 49 και ε, κανονικά πρέπει να συμφωνήσει με την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Το άρθρο 50 μας δίνει πολύ πιο ε, μεγάλη ισχύ. Γιατί όντω η ενεργειακή πολιτική είναι και αποφασιστικό μέσο και εργαλείο και αντικείμενο εξωτερική πολιτική. Ναι. Τα είπε και ο κύριο και Θέλω να σα πω ότι αύριο δεν θα ψηφίσουμε για το Ισραήλ. Με βάση την γνωμοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια μονομερή νομοδότηση, αλλά μέχρι αύριο το πρωί δεν είναι θέση να μας φέρει το κείμενο και θεωρήσαμε η εισηγήτρια και εγώ καλύτερο να αναβάλουμε αυτό το ε, θέμα ε, για να έχουμε το κείμενο στη διάθεσή μας ε, πριν αποφασίσουμε. Ελπίζω να συμφωνείτε να το αφαιρέσουμε από την αυριανή ημερήσια διάταξη και θα το βάλουμε σε επόμενη συνεδρίαση όταν θα έρθει το κείμενο της Επιτροπής. Καλό σας βράδυ, χαίρετε.